Uh, uh, Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε. Ήθελα να καθυστερήσουμε λίγο την έναρξη των εργασιών μας για να φτάσουν περισσότεροι. Φαντάζομαι ότι όλοι ευχαριστηθήκατε το χθεσινό γεύμα. Ελπίζουμε σιγά σιγά να έρχονται πάντως ε, βουλευτές όσο περνάει η ώρα. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Αλέξανδρο Δερμετσόπουλο, τον ε, πρόεδρο της ε, Επιτροπής Οικονομικών ε, Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. Ήσασταν παρόν, σχεδόν την ίδια ώρα που έφτασα και εγώ. Υπάρχουν και κάποιοι εκπρόσωποι του, των Εθνικών Κοινοβουλίων σε αυτή τη διακοινοβουλευτική συνεδρίαση που οργανώνει η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου. Ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολλή δουλειά προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε ότι σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης θα συμπεριληφθεί και θα αυξηθεί η δημοκρατική λογοδοσία και ευθύνη. Σε σχέση δηλαδή και με τα εθνικά κοινοβούλια που θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία και στις εκθέσεις επί της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης και σε ό,τι αφορά την Τραπεζική Ένωση θέλουμε να υπάρχουν διάβλη επικοινωνίας, διαβούλευσης και λογοδοσία στα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια με τον νέο μηχανισμό. Μετά από διαβουλεύσεις μαζί σας τον τελευταίο χρόνο χωρίσαμε τη συνεδρία αυτή σε δύο υποσυνεδρίες είναι ενδιαφέροντα τα θέματα, πιστεύουμε. Το ένα το έχετε αναφέρει πολύ από εσά, δηλαδή Προ ένα αποτελεσματικό σύστημα ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το δεύτερο θέμα αφορά την δημοσιονομική εξυγίνηση και τι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει, ανταλλαγή των πρακτικών δυνητικά αναμενόταν μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων. Έχουμε λοιπόν βάλει έναν κανόνα να έχουμε μόνο δίλεπτε παρεμβάσει. όταν συμπληρώσετε το καρτελάκι, το φέρνετε εδώ στο Προεδρείο και εγώ θα προσπαθήσω να διαχειριστώ το χρόνο της συζήτησης. Θα σας παρακαλώ στο καρτελάκι να αναφέρετε και τη χώρα ε, καταγωγής σας και από εκεί και πέρα είναι αυτονόητα τα πράγματα. Περνάμε λοιπόν ε, στην πρώτη συνεδρία με θέμα ένα αποτελεσματικό, ένα αποτελεσματικό σύστημα ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο πρέπει να θέσουμε τις προτεραιότητες. Ξέρουμε ότι έχουν αλλάξει πολιτικές προτεραιότητες μπορεί και να αλλάξουν ακόμη περισσότερο στο μέλλον και πολλά κράτη-μέλη θεωρούν ότι το ευρωπαϊκό επίπεδο παρεμβαίνει πλέον σχεδόν σε όλους τους τομείς της πολιτικής, στις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα προσαρμογής, ό,τι αφορά τις συστάσεις αναχώρα και τις υποχρεώσεις Πολλοί θεωρούν ότι σχεδόν επιβάλλονται, θα έλεγε κανεί, στι εθνικέ αρχέ. Συγχρόνω όμω αναγνωρίζεται ότι υπάρχει και δημοκρατικό έλλειμμα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μιλάμε δηλαδή για διακυβερνητικές συμφωνίες και κλεισμένων των θυρών ε, πάνω σε συστάσεις ε, της Κομισιόν. Και είναι πολύ δύσκολο κανείς να καταλάβει ποιος αποφασίζει για τους στόχους της πολιτικής και ποιος φέρει την ευθύνη. Θα καλωσορίσω λοιπόν τους ομιλητές μας για τη συνεδρία αυτή. Ο Φίλιπ Μαρινή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 Είναι πολύ σημαντικό να ενδιαφερθούμε για τις προοπτικές βελτίωσης του συστήματος του ΦΠΑ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο λόγος είναι ότι τα έσοδα από τον ΦΠΑ αποτελούν από δημοσιονομική άποψη πολύ σημαντική πηγή για τους δημοσιονομικούς μας πόρους. Για τη Γαλλία το ΦΠΑ αντιστοιχεί περίπου στο 50% των φορολογικών εσόδων, των καθαρών φορολογικών εσόδων ανέχεται σε περίπου 140 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2014 υπολογίζεται υπό αυτές τις συνθήκες η βελτίωση της καταπολέμησης ε, της απάτης ε, αποτελεί σημαντικό παράγοντα αυτό εφαρμόζεται ειδικότερα σε αυτό που ονομάζουμε απάτη τύπου τύπου καρουζέλ και το κοινοβουλίο μα έχει θετήσει ένα μηχανισμό ώστε οι φορολογικέ αρχές να μπορούν να πραγματοποιούν ελέγχους που τους επιτρέπουν να αμφισβητήσουν τι δραστηριότητες που επικαλείται μια επιχείρηση για να λάβει τον ενδοκινοτικό αριθμό ΦΠΑ. Αλλά θα ήθελα να αναφέρω και ένα άλλο ζήτημα, όλο και πιο σημαντικό σε θέματα ΦΠΑ είναι η ανάπτυξη των ε, πωλήσεων στο διαδίκτυο. Βάσει ενό ελέγχου που διεξήχθη τους τελευταίους μήνες από δύο συναδέλφους μου γυροσιαστές στα τελωνία του αεροδρομίου Σόλντεγκολ στο Παρίσι οι συναδελφοί μου εκπώνησαν μια ανακοίνωση στην Επιτροπή που έγινε τα έκθεση ενημερωτική διαθέσιμη στο κοινό και στο διαδίκτυο. Στην έκθεση αυτή διαβάζουμε κυρίως ότι η δράση των τελωνιακών αρχών των τελωνιακών υπηρεσιών είναι σίγουρα αποτελεσματική όσον αφορά την προστασία και την καταπολέμηση των διαφορετικών διακινήσεων, των παρεπημένων προϊόντων, των απαγορευμένων προϊόντων, όπλων, προστατευμένων ειδών, επικίνδυνων προϊόντων. Αντιθέτως όμως ε, σε φορολογικά θέματα απομένουν πολλά που πρέπει να διορθωθούν. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονό ε, ότι η έλεγχη είναι περιορισμένη... ...περιορισμένη λόγω των κανόνων που εφαρμόζονται στα... στις ταχείες αποστολές και στις ταχυδρομικές αποστολές. Όσον αφορά τις ταχείες αποστολές ε, φτάνουν τα εμπορεύματα τέσσερις ώρες πριν φύγει το αεροπλάνο. Είναι πολύ λιγότερο ακριβής η έλεγχη σε σχέση με τα παραδοσιακά εμπορεύματα. Όσον αφορά τα χειδρομικά ε, δέματα, οι υποχρεώσεις δήλωσης είναι ελάχιστες και ουσιαστικά δεν μπορούν να επαληθευτούν. Όπως γνωρίζουμε η διαδικασία δεν είναι ε, ε, μηχανογραφημένη. Συνεπώς πολλοί φόροι δεν εισπράττονται από αυτού του είδους τα εμπορεύματα. Διαπιστώνεται αυτό όταν βλέπουμε ότι στο αεροδρόμιο Ροασί τα ποσά ανέρχονται σε, σε 5,5 εκατομμύρια ευρώ έχουν, ε, δεν, ε, δεν έχουν ληφθεί ε, καθόλου χρήματα από τα ταχυδρομικά δέματα ενώ στα κανονικά εμπορεύματα 550.000. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια διαρροή του ΦΠΑ στη Γαλλία και είμαι σίγουρος και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά ο υπολογισμός των τελών εισαγωγής βασίζεται σε απλές δηλώσεις και σε ένα σύστημα το οποίο βασίζεται στην ευκολία των συναλλαγών. Αυτό ευνοεί τον κατακαιρματισμό των ε, αποστολών ε, όπως γίνεται στις online πωλήσει και είναι σαφές ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της μορφής εμπορίου διευκολύνουν ιδιαίτερα την απάτη. Έτσι λοιπόν ε, η αρχή μας βρίσκεται αδύναμη Εφόσον η ιστοσελίδα που πραγματοποιεί τι συναλλαγέ βρίσκεται στο εξωτερικό, εμεί δεν μπορούμε να προβούμε σε καμία επανόρθωση, ούτε να ασκήσουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ε, πληροφόρηση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή κοινότητα και ε, απαντάται και σε άλλους τομείς Νέου τομεί ε, που οφείλονται στην αναπτύξη της ψηφιακής τεχνολογίας. Συμπερασματικά λοιπόν θα εμείς προτείνουμε ως Επιτροπή Οικονομικών μία εισπράξη στην πηγή του ΦΠΑ εισαγωγής ε, τη στιγμή της συναλλαγής και όχι τη στιγμή άφηξης ε, των πραγματών στο τελωνίο. Οι διαμεσολαβητές των πληρωμών, οι τράπεζε, οι τοποθεσίε πληρωμών στο διαδίκτυο θα μπορούσαν να επιφορτιστούν με την εκαθάριση και τη συλλογή του φόρου αυτού. Για τις υπόλοιπες προτάσεις, επιτρέψτε μου κυρία Πρόεδρε, να ε, σας παραπέμψω στο έγγραφο το οποίο δημοσιεύτηκε από εμάς για να κλείσω. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ένα άλλο σημαντικό ζήτημα σε θέματα ΦΠΑ. Πρόκειται για την υλοποίηση της οδηγίας της 12 Φεβρουαρίου 2008. Αφορά τον ορισμό του ποσοστού ΦΠΑ που θα εφαρμόζεται στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου. Όπως γνωρίζετε, η σημαντική μεταρρύθμιση βάσει της οποίας ε, στο εξής εφαρμόζεται ο, το ΦΠΑ κατανάλωσης ε, έπρεπε να έχει εφαρμοστεί αλλά έλαβαν ε, περίοδο χάριτος το Λουξεμβούργο μέχρι το 2015 μια μεταβατική περίοδο που του ευνοεί ιδιαίτερα και που πηγαίνουμε μέχρι το 2019. Θα ήθελα να υπογραμμίσω λοιπόν ότι έχει απόλυτη προτεραιότητα η τάχιστη εφαρμογή του συμβιβασμού του 2008 για τις μεγάλες ε, κατανοητικές χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία. Κάθε χρόνο, για να μιλήσω για τη διαφορά ποσοστού μεταξύ του ΦΠΑ όπου βρίσκεται μια πλατφόρμα και το κράτος κατανάλωσης μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ που λείπουν. Κυρία Πρόεδρε, έχω ολοκληρώσει. Θέλω να υπενθυμίσω τέλος ότι η Επιτροπή μας το Δεκέμβριο διατήρησε επιφύλαξη όσον αφορά την οδηγία για μια τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ εκτεταμένο και δεν μπορεί κανείς να το εξετάσει μέσα σε πέντε λεπτά γιατί το έκανα και εγώ, το εξέτασα, το παρουσίασα την πρόσφατα. Τώρα λοιπόν θα περάσουμε στον εκπρόσωπο του ε, Δανέζικου Κοινοβουλίου, τον κύριο Γένσεν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, πρόσκληση ε, και που μου δίνει τη δυνατότητα να σας ε, ενημερώσω για το πώς ακριβώς εφαρμόζουμε το ΦΠΑ στη Δανία και πώς αποφεύγουμε την αποφυγή καταβολής του ΦΠΑ στη χώρα μου. Το 20% των φορολογικών εσόδων στη Δανία είναι από το ΦΠΑ. Και μπορώ να σα εξηγήσω πάρα πολύ καλά πώ λειτουργεί το σύστημα στη Δανία. Εμείς έχουμε δύο συντελεστέ, έναν 25% και έναν μηδενικό συντελεστή για το ΦΠΑ. Το 25% ισχύει για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Και υπάρχουν μόνο ελάχιστες εξαιρέσεις, ε, παραδείγματο χάρη, οι εφημερίδε, ε, οι χρηματοψηφιακές υπηρεσίε. Ε, και τα ενίκια εξαιρούνται. Τώρα, ΦΠΑ καταβάλουν ε, στη Δανία όλοι οι επιτιδευματίες ε, που εργάζονται οι οποίοι οποτεδήποτε προσφέρουν τις υπηρεσίες τους επιβάλλουν και ένα ΦΠΑ 25% μέσα σε 12 μήνες ε, και μια επιχείρηση εφόσον πλώνει πάνω από 6.500 ευρώ πρέπει να καταβάλει ΦΠΑ, γίνεται ένας ε, συμψηφισμός και το ΦΠΑ που έχει καταβληθεί ε, μπορεί κανείς να το αφαιρέσει από τους ε, καταβαλόμενους φόρους. Ας δούμε λιγάκι ποιο είναι το κενό. Έχουμε λοιπόν μεγάλη πίεση στους προϋπολογισμούς, αλλά το κενό, το, η τρύπα από το ΦΠΑ είναι πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή 2,7% για το 2010. Αυτό είναι το ποσοστό που αντιστοιχεί στο μη, στο μη καταβληθέντα φόρο για το 2010. Μιλάμε όμως για 13 δις ευρώ που εισπράχτηκαν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στην ε, Δανία έλεγξε αυτό το κενό ε, λόγω μη καταβολή σε ΦΠΑ, καθαρά θεωρητικά βέβαια. Και στη Δανία αντιστοιχεί το 10%, κάτι που είναι ένας, ένα αρκετά χαμηλό ποσοστό σε σχέση με άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τομέας λοιπόν του ΦΠΑ παρουσιάζει μια ικανοποιητική εικόνα ικανοποιητική είναι η κατάσταση για το πώς ακριβώς αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες και οι πολίτες στο ΦΠΑ στη Δανία. Οι περισσότεροι πολίτες καταβάλουν το φόρο που τους αναλογεί χωρίς να διαματήρονται, χωρίς να εξαπατούν. Ξέρετε γιατί, διότι για τους φόρους που καταβάλουν έχουν υψηλό ανταποδοτικό επίπεδο. Βεβαίως και παρισφρίουν λάθη και βεβαίως και υπάρχουν κάποιες μικρές απάτες. Παρότι λοιπόν το σύστημά μας του ΦΠΑ είναι τόσο απλό και παρότι η προθυμία είναι μεγάλη, όπως σας είπα, παρισφρίουν λάθη και υπάρχουν και περιπτώσεις απάτης. Κάθε χρόνο εφαρμόζουμε μία έρευνα, μία μελέτη συμβατότητας και εκεί ε, διαπιστώνουμε ε, το, ότι πράγματι οι Δανείοι είναι ιδιαίτερα συμμορφωμένοι με το σύστημά τους. Ε, στην έρευνα αυτή διαπιστώνουμε επίσης πού μπορούν να παρισφρήσουν λάθη. Διαπιστώσαμε ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα υπάρχουν στις οικογενειακές επιχειρήσεις με ένα ή δύο απασχολούμενους. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις παρουσιάζουν λιγότερα προβλήματα. Έτσι λοιπόν σε αυτές τις οικογενειακές επιχειρήσεις χωρίς υπαλλήλους το κενό είναι στο 13% με εταιρείε από 1 μέχρι 12 ε, υπαλλήλους το κοινό ε, προσδιορίζεται στο 3% και σε επιχειρήσεις άνω του 12 υπαλλήλων είμαστε στο 0,6%. Βεβαίως πρέπει να γνωρίζουμε ποιες επιχειρήσεις πρέπει να ελεγχθούν οποτεδήποτε ασχολούμεθα με την ίσπραξη του ΦΠΑ. Τα μεγαλύτερα λάθη ε, που εντοπίζονται σε επιχειρήσεις αφορούν το ότι καταβάλλεται μικρότερο ΦΠΑ από αυτό που αναφέρεται στα λογιστικά βιβλία. Και πολλές φορές ε, ε, δεν είναι δεν είναι σωστή η τεκμηρίωση, τα έγγραφα δηλαδή που συνοδεύουν το ΦΠΑ. Αυτά είναι τα βασικά αίτια. Στην ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, προσπαθούμε να εντοπίσουμε το γιατί ακριβώς προκύπτουν αυτά τα κενά ε, ΦΠΑ στα κράτη-μέλη και γιατί το κενό αυτό είναι τόσο μικρό στη Δανία. Από τη δεκαετία του 60 υπάρχει αυτό το σύστημα ΦΠΑ στη Δανία και εμείς ε, δεν προβήκαμε σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Απλά κατά καιρού ε, προσαρμόζαμε το ΦΠΑ οποτεδήποτε εντοπίζαμε ότι υπάρχουν προβλήματα, οποτεδήποτε εντοπίζαμε το ότι οι επιχειρήσεις είχαν πρόβλημα πρόβλημα κατανόησης ε, των ε, διατάξεων. Κάθε χρόνο λοιπόν ε, εκτελούμε κάποια προγράμματα με την έννοια ότι οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών επισκέπτονται τους υποκείμενους σε φόρο και συζητούν μαζί τους για να διορθώσουν ενδεχόμενα λάθη. Η έρευνα, η μελέτη αυτή συμβατότητας γίνεται σε 3.000 επιχειρήσεις που επιλέγονται κάθε φορά και με τον τρόπο αυτό γίνεται ενδελεχής ανάλυση του ΦΠΑ. Αν λοιπόν κάτι εντοπιστεί ότι δεν είναι σωστό, παρεμβαίνουν οι υπηρεσίες και διορθώνουν τα λάθη. Και επίσης καταγράφουν τι είδους λάθη προκύπτουν. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι μπορούμε σιγά σιγά να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και κάθε χρόνο να καταβάλει το ΦΠΑ χωρίς λάθη. Όσον αφορά τώρα την έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκεί δεν αναφέρεται γιατί το κενό από την εισπραξή του ΦΠΑ είναι τόσο μικρό, παρότι σε εμά η πίεση ε, καταβολής ΦΠΑ είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Εκτός λοιπόν από την προθυμία καταβολής υπάρχει και κάτι άλλο. Η κατα Γραφή των επιχειρήσεων είναι ουσιαστική. Έχουμε ένα κεντρικό μητρό, πολύ καλά ε, διαρθρωμένο και υπάρχει και μια άλλη εξέλιξη, ότι σε εμά οι ε, συνδιαλλαγές υποκείμενες στο ΦΠΑ είναι ψηφιοποιημένες. Και ίσως ε, το κενό, το ότι είναι μικρό, να οφείλεται και στο ότι εμείς έχουμε ένα απλό σύστημα καταπολής ΦΠΑ. Σας είπα μόνο δύο συντελεστές, ο ένας του 25% και ο άλλος μηδενικός συντελεστής. Υπάρχει λοιπόν αυτό το μικρό κενό εισπράξεων και κάθε χρόνο προσπαθούμε να το περιορίσουμε, το καταφέρνουμε και εμείς ε, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και κάποια φαινόμενα του σειρμού που είναι απάτε σε σχέση με το ΦΠΑ, φαινόμενα καρουσέλ επίσης όπως λέγονται. Στην ε, Δανία υπάρχει θετική ε, αντιμετώπιση απέναντι στα ευρωπαϊκά μέτρα γιατί οι επιχειρήσεις είναι αναγκασμένες να συνεργάζονται και να καταπολεμούν την απάτη με θέματα ΦΠΑ. Γι' αυτό λοιπόν εμείς προσπαθούμε να εφαρμόζουμε το συντομότερο δυνατόν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά είχα να σας πω για το ΦΠΑ στη Δανία. Ευχαριστώ. Είμαι κάπως γενναιόδορη με το χρόνο. Ε, μπορούμε να επανέλθουμε μετά. Μέχρι στιγμής ε, είναι ένας μόνο μιλητής που έχει εγγραφεί στον κατάλογο, γι' αυτό είμαι γενναιόδορη. Όποιοι έρχονται σιγά σιγά ενδεχομένως θα μπορούν να προσθέσουν στον κατάλογο αυτό. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Γιάννους Βέρης από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2011 όταν δημοσίευσε την ανακοίνωσή της για το μέλλον του ΦΠΑ μίλησε για ένα ανανεωμένο σύστημα ΦΠΑ και περιέγραφε εκεί τα βασικά αιτήματα και τα βασικά σημεία ενός τέτοιου συστήματος. Καταρχάς, να σχολιάσω το σύστημα ΦΠΑ γιατί μιλάμε ένα ενιαίο σύστημα δήλωσης. Αν δείτε τι προτείνεται το 2013 στις 15 Νοεμβρίου στο ΕΚΟΦΗΝ υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσον η νέα πρόταση οδηγεί σε απλούστευση. Αν δείτε δηλαδή τη συχνότητα των δηλώσεων και τις προθεσμίες καταβολής του ΦΠΑ θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει κίνδυνος να έχουμε αρνητικό αντίκτυπο στις ταμιακές ροές. Το δεύτερο σημείο το οποίο θεωρώ ότι είναι σημαντικό αν θέλουμε να έχουμε ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα ΦΠΑ είναι ότι αν υπάρχουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και ενιαία δέσμη κανόνων, αυτό θα είναι θετικό. Ο γερουσιαστής Μαρινή είπε ε, πράγματα που τα θεωρώ πολύ σωστά. Πολλά κράτη-μέλη θεωρούν ότι ε, πρέπει να έχουν αυτά τα δικά του συστήματα για τους μειωμένους συντελεστές. Τα τελευταία δέκα χρόνια πολύ βιώσαμε αυτό το φαινόμενο, ότι κάποια κράτη δηλαδή εντάσσουν συστηματικά ε, κάποιες διατάξεις στα συστήματά τους. Εάν δεν αλλάξει η κατάσταση στα κρατημέλη, αυτό το εμπόδιο θα συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια. Αν θέλουμε να έχουμε ένα ισχυρότερο σύστημα ΦΠΑ, θα πρέπει επίσης να καταπολεμήσουμε την απάτη. και θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικό το σύστημα του ΦΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να πω ότι αν δείτε τα συνολικά έσοδα από το ΦΠΑ στην Ένωση δεν είναι τόσο υψηλά. Θέλουμε να τα αυξήσουμε. Και σε ό,τι αφορά τα έσοδα που δεν φτάνουν στον προπολογισμό, αυτά έρχονται σε ένα 12%. Όταν προσχωρήσαμε το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χάσαμε το 10% των εσόδων μας από το ΦΠΑ. Το ίδιο συνέβη και στα άλλα κράτη τα οποία προσχώρησαν εκείνη την εποχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε ένα ρόλο και η κατάργηση κάποιων τελωνιακών ελέγχων Έχουμε επίσης τη λεγόμενη απάτη τύπου καρουσέλ, την αλυσιδωτή απάτη περί τις επιστροφές. Και αυτό το φαινόμενο ε, βλέπουμε να εξαπλώνεται. Πρέπει να το περιορίσουμε, πρέπει να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές. Με βάση λοιπόν την εμπειρία μας των τελευταίων ετών, διαπιστώσαμε ότι οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες για τις φορολογικές βάσεις. Σε όλα τα κράτη-μέλη Υπάρχουν παράμετροι, υπάρχουν σχετικές παράμετροι, τα σχετικά εργαλεία. Θέλουμε λοιπόν να είναι πιο γρήγορη και ομαλή η πρόσβαση στην ενημέρωση της πληροφορίας για να μπορέσουμε να διευρύνουμε ακόμη περισσότερο την διακρατική συνεργασία. Και επειδή υπάρχουν κάποια προϊόντα που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις απάτες, ναι, μεν πρέπει να ανταλλάξουμε τι προσεγγίσεις μα και τι πρακτικέ μα, αλλά να προχωρήσουμε και στι απαραίτητε βελτιώσει. Αν δηλαδή βλέπουμε ξαφνικές, σοβαρές απάτες σε επίπεδο κάποιου κρατου. θα πρέπει να έχουμε έναν μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης που θα τίθεται σε ισχύ. Είχαμε και κάποιες πρωτοβουλίες στην Ουγγαρία κατά το παρελθόν θα μπορούσαν να δουν τα άλλα κράτη-μέλη τι κάνουμε εμείς στη χώρα μας. Επίσης βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλες δέσμες, παρτίδες προϊόντων που πολλούνται, τα παλιοσίδερα, τα απορροκυπευτικά προϊόντα ε, κρέατος, όλα αυτά. Πώς διακινούνται, πώς πολλούνται. Βλέπουμε την απάτη να εξαπλώνεται και να καλύπτει μια ευρύτερη γκάμα από προϊόντα. Για τα παλιοσίδερα, για κάποια δημητριακά, προϊόντα από σιτηρά δημητριακά, κάναμε κάποιες κινήσεις που μας επέτρεψαν να περιορίσουμε την απάτη. η καταπολέμηση απάτης μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική αν επιβληθούν ε, και οι ψηλότεροι συντελεστέ. Κάποιες φορές βλέπουμε να μην υπάρχει μετακίνηση του προϊόντος από ένα κράτος μέλος στο άλλο, αλλά μετακίνηση κάποιου εγγράφου από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Και έτσι γίνεται η απάτη. Πρέπει λοιπόν να ερευνώνται πολύ καλύτερα και τα ε, εμπορεύματα και τα φορτηγά, αλλά ακόμα περισσότερο πρέπει να ελέγχονται τα έγγραφα. Γιατί όπως είπα εκεί πολλές φορές εντοπίζεται η απάτη. Θα πρέπει να παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά όλες αυτές τις μετακινήσεις προϊόντων και εγγράφων. Ευχαριστούμε πολύ. Έχω ακόμα περιθώριο για έναν ομιλήτη. Έχω τώρα τον Τέντορο Στοϊάν, ένα από του αντιπροεδρού της Επιτροπής Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπόλς. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το σημερινό σύστημα ΦΠΑ όταν εισήχθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ονομαζόταν μεταβατικό σύστημα και έχει παραμείνει μεταβατικό προσωρινό εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα καταφέρουμε να μετακινηθούμε από την αρχή του προορισμού στην αρχή της προέλευσης στις καταβολές του ΦΠΑ. Ωστόσο δεν πιστεύω ότι κάτι τέτοιο πρόκειται να το δούμε μέσα στα επόμενα χρόνια. Εμείς ε, λοιπόν μόλις εγκρίναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε επίπεδο Συμβουλίου ένα πολύ ισχυρό μηχανισμό καταπολέμησης της ε, αποφυγής ΦΠΑ και όχι μόνο της αποφυγής ΦΠΑ και ε, της απάτης ΦΠΑ είναι το σε 2014 2014-2020. Το Φισκάλι, λοιπόν, το πρόγραμμα Φισκάλι αποτελείται από δύο κυρία τμήματα. Το πρώτο αφορά την οικοδόμηση και την αναβάθμιση των ε, πληροφοριακών συστημάτων, ενός συστήματος ενημέρωσης εστιασμένου στην επικοινωνία μεταξύ Υπουργείων Οικονομικών όλων των κρατών μελών. Το δεύτερο κομμάτι αυτού του προγράμματος φυσκάλης το οποίο αν δεν κάνω λάθος ε, δεν χρησιμοποιείται επαρκώς είναι η ανταλλαγή εμπειριών σε επίπεδο προσωπικού και προσωπικού υψηλού επίπεδου των Υπουργείων Οικονομικών των κρατών μελών με στόχο την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών αναχέτησης της ε, φοροαποφυγής, ε, της ε, φοροδιαφυγής και ούτω καθεξής. Πιστεύω ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να εστιαστούν σε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί, διότι αυτό το πρόγραμμα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην εκπλήρωση των στόχων μας, δηλαδή της αναχέτησης αυτών των κακών συνηθιών που δυστυχώς λαμβάνουν χώρα στα κράτη-μέλη μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ήμουν λίγο αυστηρή με τους ομιλητές μου γιατί νόμιζα ότι θα είχαμε πάρα πολλές κάρτες ε, πλημμυρολόκληρη αλλά έχω μόνο άλλον ένα ομιλητή και μετά θα περάσουμε στους συμμετέχοντες στο πάνελ από το Κοινοβούλιο της Πολωνίας λοιπόν ο Ντάριος Ριζάτη πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Οικονομικών και που υπήρξε παλαιότερα ευρωβουλευτής. Παρακαλώ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Το σύστημα ΦΠΑ συχνά αποτελεί το αντικείμενο κατάχρησης και απάτης. Δεν μπορώ παρά να υποστηρίξω τα επικριτικά σχόλια των προλαλήσαντων στην Πολωνία η κλίμακα της απάτης ανέχεται στο 10 με 15% όλων των φορολογικών εσόδων ε, για τον προπολογισμό. 4 με 7% όλων των ε, δημοσιονομικών εσόδων. Μιλάμε για μια τεράστια τρύπα στα δημόσια οικονομικά που παρενοχλεί και διαστρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Ουσιαστικά σημαίνει ότι κάποιες επιχειρήσεις έχουν πλεονεκτική θέση Απλά και μόνο διότι ε, πραγματοποιούν απάτη. Έχουμε αυτό το σύστημα το καρουζέλ, ε, ψευδείς ε, συναλλαγές λαμβάνουν χώρα και μετά καθαρίζονται και συχνά έχουμε τέτοιες επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν μία συναλλαγή και μετά εξαφανίζονται, πηγαίνουν και δημιουργούν έδρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα σε καύσιμα όπως μέταλλα και καύσιμα αυτή η απάτη είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Είναι πολύ δύσκολο να καταπολεμήσει κανεί αυτού του είδου την απάτη. Πρέπει να συντονίσουμε τι προσπαθίε μα σε και Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πιστεύω κάποιοι τρόποι καταπολέμησης αυτού του είδου ε, του εγκλήματος, το έγκλημα, το αντίστροφο ΦΠΑ, η αντίστροφη. της ουσιαστικά στα προϊόντα μετάλλων ε, μπορεί να βοηθήσει σε τεράστια μείωση της απάτης. Έτσι συνέβη με, όταν ελήφθη αυτή η απόφαση. Επίσης πρέπει να έχουμε καλή επικοινωνία μεταξύ μας για τις ε, συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα. Όταν ε, εκδίδεται ένα τιμολόγιο θα πρέπει κάποιος να ειδοποιεί τη φορολογική του, την εφορία του και μετά το, όλο το δίκτυο των εφοριών θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να καταπολεμήσει την απάτη. Επίσης πρέπει να καταχωρούμε σε μητρότητες επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους εμπόριο. Έχουμε και κάποια εξαιρετικά παραδείγματα από την τσεχική δημοκρατία. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τσέχοι συνάδελφοι εδώ στην αίθουσα. Θα μπορούσαν ίσω να μοιραστούν μαζί μα ε, τι δικέ του εμπειρίε ε, επί του θέματο. Θα μπορούσαν να αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμο για όλου μα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαρίνη, επιθυμείτε να κάνετε κάποια άλλα σχόλια. Ξέρω ότι έχετε αρκετά να πείτε ακόμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν δει κανεί ε, τα αποτελέσματα του ελέγχου που κάναμε στη Γαλλία σε ό,τι αφορά το εμπόριο online, το ηλεκτρονικό εμπόριο, βλέπει κάποια πράγματα και αυτό το ανέφερα ουσιαστικά απευθυνόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι για να προχωρήσουμε στο θέμα του ελέγχου και για να μειώσουμε τις διαρροές από έσοδα ΦΠΑ, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενταχθούμε στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου. Αυτές είναι οι δύο βασικές προτάσεις μας λοιπόν. Πρώτον, η καθιέρωση ενός συστήματος αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ τελωνίων ε, και ενδιάμεσων στο, των ταχυδρομικών αποστολών ε, και αποστολών εμπορευμάτων, φορτίων κτλ. Και, πρώτη, και δεύτερη μάλλον πρόταση, εισαγωγή ε, ενός φόρου παρακάτω στην πηγή που καταβάλλεται δηλαδή τη στιγμή της συναλλαγής και όχι όταν φτάσει το προϊόν το εμπόρευμα στο τελωνίο και ενδιάμεσα προβαίνουν στην εκαθάριση και στην ίσπραξη του φόρου. Τις, υπογρα... τις ε, υπογραμμίζω τις προτάσεις αυτές γιατί φυσικά ε, ίσως να μην μπορεί ένα κράτος να εφαρμόσει τις διατάξεις αυτές αν δεν είναι σύμμορφες με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο. Θα πρέπει λοιπόν κύριε Πρόεδρε πιστεύω να συζητηθούν, να τεθούν σε συζήτηση όλες αυτές οι προτάσεις. Επειδή είναι και πολύ μεγάλη οικονομική σημασία του κλάδου αυτού. Επίσης, οι πωλήσει εξ αποστάσεως στη Γαλλία είναι μια δραστηριότητα αυτή που ουσιαστικά αφορά πάνω από δύο στους τρεις Γάλλους. Και ο ετήσιος κύκλος εργασιών του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι της τάξης των 45 εκατομμυρίων σε ό,τι αφορά τα υλικά αγαθά, 25 δισεκατομμύρια ευρώ ο τζίρος από τις εξαποστάσεις πωλήσει. Αν λοιπόν δεν μπορέσουμε να οργανωθούμε για να προσαρμόσουμε την νομοθεσία και τις διαδικασίες μας, είναι σαφές ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι άλλο θέλουμε, αλλά θα υπονομεύσει τα έσοδα από τα φορολογικά μας έσοδα η τεχνολογία, η τεχνολογική πρόοδος. Άρα θα μειωθούν τα φορολογικά έσοδα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν γέννη. Um, Μάλιστα, κατάλαβα. Και ως Μπενέση, ή κάπως έτσι θέλει να λάβει τώρα το λόγο. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ε, φαντάζομαι σήμερα μπορώ να μιλήσω τσέχικα στη γλώσσα μου και θα ήθελα να τοποθετηθώ σε αυτά που είπε ο συνάδελφος από το Πολωνικό Κοινοβούλιο που είπε ότι ε, καλό θα ήταν ε, να τοποθετηθεί και ένας Τσέχος. Κοιτάξτε, εγώ είμαι πρόεδρος ε, της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και δεν είμαι απαραίτητα επαΐων των θεμάτων ΦΠΑ στην Τσεχία. Αλλά Παρ' όλα αυτά μπορώ να διαβεβαιώσω τον Πολωνό συνάδελφο ότι η νέα κυβέρνηση στην Τσεχία που μόλις ε, ανέλαβε την εξουσία της χώρας, η νέα λοιπόν κυβέρνηση επιθυμεί διακαώς να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την ε, φοροαπάτη ε, και την φοροδιαφυγή κυρίως σε επίπεδο ΦΠΑ και σε σχέση με τα αλκοολούχα ποτά. Ήδη ε, έχουμε επιτύχει σημαντικά στην απάτη ΦΠΑ ως προς τα καταναλωτικά αγαθά. Άρα δηλαδή είμαστε στην ευτυχή θέση να μπορούμε να πούμε ότι ξεκίνησε αποτελεσματικά ο αγώνας μας. Έχουμε ήδη σημειώσει κάποια επιτυχία και ελπίζω ότι θα βελτιωθούμε περαιτέρω. Σας ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω κάποιες ε, ερωτήσεις ε, προς την Επιτροπή. Ίσως λοιπόν η Επιτροπή μπορεί να προετοιμαστεί και μετά να λάβει το λόγο και να απαντήσει. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Γιάννος Βέρος, ο οποίος έχει και αυτός να κάνει κάποια σχόλια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με την πρόταση του Γερουσιαστού. Δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τις συναλλαγές στο διαδίκτυο. Πρέπει να εξετάσουμε γενικότερα όλες τις αυτόματες ε, συναλλαγές ε, μεταξύ κρατών μελών ε, και αρχών τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία που έχουν αποθηκευτεί σε άλλα κράτη-μέλη σε σχέση με το ΦΠΑ. Πιστεύω καθίσταται σαφές ε, ότι τα υπολογιστικά συστήματα των κρατών μελών περιέχουν πολύ περισσότερα δεδομένα από όσα ανταλλάσσονται ε, μεταξύ των κρατών μελών πολύ λιγότερα δηλαδή δεδομένα διαθέσιμα για άλλα κράτη-μέλη. Θέλω να το πω σε αυτό στον Πολωνό συνάδελφο, γιατί και εγώ έχω την ίδια εμπειρία στην Ουγγαρία. Το ίδιο συμβαίνει και στη χώρα μα όπω και αυτό που μα περιγράψετε εσεί. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, πιστεύω, να προβούμε σε μια κοινή αξιολόγηση των εμπειρία των αντίστροφων χρεώσεων. Αυτό το σύστημα των αντίστροφων χρεώσεων, το reverse charge, θα μπορούσαμε πούμε, να το εξετάσουμε σε πολωνικό και ουγγρικό πλαίσιο και να εισάγουμε δηλαδή τις ίδιες χρεώσεις στην ίδια κατηγορία προϊόντων και να δούμε από κοινού ποια ήταν τα αποτελέσματα της εισαγωγής αυτής της μεθόδου, για παράδειγμα στα προϊόντα μετάλλων ε, και να δούμε τι συνέβη στην Ουγγρία, τι συνέβη στην Πολωνία και να δούμε και τι συνέβη σε θέματα απάτης, ε, διότι μπορεί η απάτη να ξεκινήσει από τέτοια προϊόντα, αλλά μπορεί να μετακινήθηκε μετά σε άλλα προϊόντα. Αξίζει πιστεύω λοιπόν τον κόπο να εξετάσουμε μια τέτοια κατηγορία προϊόντων και με αυτή την πρακτική και αυτή η πρακτική μάλιστα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί γενικότερα, να επεκταθεί και σε άλλε χώρε και σε άλλου τομεί. Ε, πρέπει να δούμε όλου του τους ε, στην αγορά Όταν μιλάμε για μεμονωμένους επιχειρηματίες, για επιχειρήσεις, πρέπει να δούμε και το πώς μπαίνουν στην αγορά. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν με ε, σύγκριση των εμπειριών στα διάφορα κράτη-μέλη πριν προβούμε σε νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόεδρος, ναι, όπως ανέφερα προηγουμένως στο τελευταίο κοινοβούλιο είχα εκπονήσει μια έκθεση που διερευνούσε πολλές από αυτές τις επιλογές γιατί πολλά κράτη-μέλη ε, χρησιμοποιούν αυτούς τους μηχανισμούς reverse charge αντίστροφης χρέωσης για κάποια ε, υλικά και αγαθά ιδιαίτερης ευαισθησίας. Ε, είναι δύσκολο φυσικά να εφαρμοστούν στα πάντα, αλλά εγώ αναρωτιόμουν στο πλαίσιο των απατών τύπου καρουζέλ, αυτό το γαϊτανάκι. Τώρα που έχουμε τόσα πολλά συστήματα μηχανογραφημένα και έχουμε την ανάγκη ανταλλαγή πληροφοριών Μπορεί κάπως ε, να ξεφύγει κάποιος από αυτή την εξαίρεση, τη διασυνοριακή. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες ε, μεταφορές κεφαλαίων που, χρημάτων που πρέπει να παρακολουθούνται διασυνοριακά. Δεν υπάρχει αυτή η τεχνολογία για να καλύψει αυτό το παραθυράκι. Διότι, αν θυμηθούμε τα όσα ανέφερε ο Γάλλος συνάδελφος ε, με τα, τα θέματα για τα εμπορεύματα, Εάν αρχίσουν να γίνονται υπερβολικά αδιάκριτες οι υπερβολικές, οι τελωνιακές επιθεωρήσεις, τότε θα έχουμε πρόβλημα όσον αφορά την ελεύθερη διακίνηση, την ελεύθερη κυκλοφορία που αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη μας δικαιώματα. Τι θα κάνουμε, θα το παρακολύσουμε ώστε να ε, εισπράττουμε το σωστό ποσοφόρον. Επιτροπή, θα μπορούσατε να μα πείτε κατά πόσο μπορείτε να απαντήσετε σε κάποια από αυτά τα προβλήματα. Έχουμε αρκετό χρόνο. Η επόμενη συζήτηση δεν θα αρχίσει πριν τι 14, οπότε αν θέλει οποιοδήποτε να μιλήσει, παρακαλώ στείλτε μια κάρτα ή ε, σηκώστε χέρι σας για να σας ε, δούμε. Ε, Merci, Madame ε, la Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να δώσω κάποιες απαντήσεις. Σε αυτή την ψηφιακή οικονομία, καταρχάς, η οποία έχει δύο κλάδους. Νομίζω ότι ο γερουσιαστής Μαρινή το ανέφερε. Ο πρώτος κλάδος είναι η παραγγελία αγαθών από το διαδίκτυο και μετά η παράδοση αυτών. Έχουμε τι εξαποστάσεω πωλήσει, εκεί έχουμε πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα έλεγχο από τα κράτη-μέλη και τα εμπορεύματα που προέρχονται από τι τρίτε χώρε. Εκεί με την ευθύνη των τελωνικών υπηρεσιών πρέπει να ελέγχεται η άφηξη των εμπορεύματων αυτών. Και βέβαια οι τελωνιακοί πολύ δύσκολα μπορούν τι μικρέ αποστολέ, όπω τι λέμε, να τι ελέγξουν, εφόσον υπάρχουν εκατομμύρια τέτοιε αποστολέ ε, ημερησίως. Έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε στην Κομισιόν πριν από ένα με δύο μήνες μία μελέτη και περιμένουμε τα αποτελέσματα περί τα μέσα αυτής της χρονιάς για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από νομοθετικής πλευράς. Και αυτό κυρίω επειδή είδαμε ότι υπάρχει σημαντική απάτη. Εταιρείε οι οποίε εγκαθίστανται σε μια τρίτη χώρα και αποστέλουν δέματα χαμηλή αξία ε, μέσα στην απαλλαγή Έχουμε μια απαλλαγή 10 έως 22 ΦΠΑ, κάποια δηλαδή CD ή DVD που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομίμως, γιατί απαλλάσσονται εάν είναι κάτω από μια συγκεκριμένη τιμή. Και δεν ξέρουμε πώς θα έπρεπε να το καταργήσουμε αυτό. Από την άλλη πλευρά, αν καταργήσουμε αυτή την απαλλαγή, πώς μετά μπορούμε να ελέγχουμε. Ο γερουσιαστής Μαρινή ανέφερε κάποιες προτάσεις, εμείς ε, θα εξετάσουμε, βέβαια υπάρχει στην πηγή. Μπορεί να είναι μια λύση, αλλά απαιτεί συνεργασία ιδίως με τρίτες χώρες ή με μεσάζοντες για την ίσπραξη του ΦΠΑ. Και αυτό μας δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Δεύτερο, δεύτερος κλάδος της ψηφιακής οικονομίας είναι οι λεγόμενες ψηφιακές υπηρεσίες. Δηλαδή, όταν κάποιος κατεβάζει, μεταφορτώνει κάποια προγράμματα ηλεκτρονικά ηλεκτρονικές υπηρεσίες, broadcasting κτλ. Από την 1η Ιανουαρίου του 2015 θα ισχύσει ένας κανόνας φορολόγησης στη χώρα διαμονής του καταναλωτή. Είχαμε μια μεταβατική περίοδο από το 2008, ε, επταετής, αρκετά δηλαδή μακροχρόνια μεταβατική περίοδος, το Λουξεμβούργο ήθελε να προστατεύσει τα φορολογικά του έσοδα Ξέρετε ότι στην ψηφιακή οικονομία ένα δις είναι τα, έξοδα, τα έσοδα, συγγνώμη, τα φορολογικά του Λουξεμβούργου. Θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια μονοαπευθυντική μήνυ θηρίδα, για πρώτη φορά δηλαδή στην ιστορία του ΦΠΑ, ένα κράτος μέλος μπορεί να εισπράττει ΦΠΑ για ένα άλλο κράτος μέλος. Δηλαδή το κράτος μέλος όπου είναι κατεστημένος ο πολιτής, εισπράττει το ΦΠΑ για το κράτος μέλος όπου είναι κατεστημένος τελικός καταναλωτής. Και αυτό γίνεται σε κοινοτικό επίπεδο για πρώτη φορά στην ιστορία. Όμως, τίθεται το εξή θέμα. Τι γίνεται με τα τρίτα κράτη. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα σύστημα ενιαία στηρίδα για τις τρίτες χώρες που είναι όμως εθελοντικό. Και διαπιστώσαμε ότι πολύ λίγε είναι οι εταιρείε που έχουν εγγραφεί σε αυτό το εθελοντικό σύστημα. Άρα έχουμε μεγάλη φοροδιαφυγή από τις τρίτες χώρες ή από πολιτέ που είναι κατεστημένοι σε τρίτε χώρε και οι οποίοι παρέχουν ηλεκτρονικέ υπηρεσίε χωρί να πληρώνουν τον κοινοτικό ΦΠΑ. Και εδώ θα ξεκινήσουμε με την κατάρτιση ενός, ε, μιας εντολής διαπραγμάτευσης, θα την υποβάλουμε στο Συμβούλιο ώστε να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις με τις τρίτες χώρες και κυρίως βέβαια τους βασικούς μας εταίρους, τους βασικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά σε ό,τι αφορά την ψηφιακή οικονομία. Ένα άλλο ζήτημα. Συνεργασία και απάτη. Έγινε πρόοδος. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν τα νομικά μέσα και εργαλεία για να, απο, να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά ε, την φορολογική απάτη. Είναι τοπικό να θεωρεί κανείς ότι ένα κράτος μόνο του μπορεί ε, να καταπολεμήσει αποτελεσματικά την ΑΠΑΤ. Χρειάζεται διασυνοριακή συνεργασία. Νομικά μέσα και εργαλεία υπάρχουν. Αλλά πού είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει επαρκή βούληση από πλευρά κατών μέλων για συνεργασία. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Έχουμε το Eurofisk, μια δομή που επιτρέπει την πιο ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μέλων. Δεν λειτουργεί όμω τόσο καλά όσο θα θέλαμε ή όσο είχαμε νομίσει στην αρχή. Εξού και πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία. Υπάρχει όμω μια πρωταρχική ευθύνη που είναι ε, για τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τα εργαλεία που του παρέχει η Κομισιόν. Το reverse charge, αυτή η αντιστροφή τη επιβάρυνση το, το λικιντασιό, αυτή η κυκλική απάτη, η απάτη τύπου καρουσέλ. Δεν αφορά μόνο τις ενδοκινοτικές συναλλαγές. Υπάρχουν και εσωτερικές συναλλαγές που γίνονται με εξαφανισμένους εμπόρους κτλ. Εκεί έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις. Νομίζω στηρίζονται αυτές και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Και θέλουμε να δούμε τη φορολόγηση των ενδοκινοτικών συναλλαγών, να την επανεξετάσουμε, να θεωρήσουμε. Και ίσω η αστροφή τη επιβάρυνση, το reverse charge, θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικό μέτρο. Δεν είναι πανάκια όμω, γιατί αυτό το σύστημα προκαλεί άλλα προβλήματα, δηλαδή μεταφέρει την ίσπραξη του ΦΠΑ στο στάδιο κοντά στην τελική κατανάλωση. Άρα, μία πρόσθετη δυσκολία για τη φορολογική διοίκηση σε ό,τι αφορά την ίσπραξη του ΦΠΑ. Έχουμε το παράδειγμα των είπα, που έχουν ένα φόρο πωλήσεων, το sales tax, φόρο πάνω στο τελικό, στην τελική πώληση. Εδώ έχουμε όμως ποσοστά απάτης της τάξης 30 έως 40%. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το sales tax το αμερικανικό πιο αποτελεσματικό από το ΦΠΑ. Συνεργαζόμαστε αυτή την περίοδο με τα κράτη μέλη και με μια ομάδα 40 εμπειρογνωμόνων που παρέχουν συμβουλές στην Κομισιόν και εξετάζουμε τρεις πιθανές λύσεις. Το σύστημα ΦΠΑ όμως, το κοινοτικό σύστημα το οποίο εγκρίναμε το 1979, πάνω από 40 χρόνια πριν, έχει απαρχιωθεί. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη φύση της σημερινής οικονομικής δραστηριότητας, τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται επιχειρήσεις και θα πρέπει και την ηλεκτρονική διοίκηση να τη συμπεριλάβουμε. Όμως δεν το έχουμε πράξει ακόμη σε σχέση και σε σύγκριση με τρίτες χώρες ή στερούμε, υπολοιπόμαστε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε επίση ένα σύστημα ΦΠΑ που ενέκριναν το 67, εξι κράτη-μέλη. Και για να μεταρρυθμιστεί αυτό το σύστημα 50 χρόνια μετά, πρέπει να συμφωνήσουν 28 κράτη-μέλη. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Εμείς θα υποβάλουμε προτάσεις και το κάνουμε σε επίπεδο Συμβουλίου. Υπάρχουν βέβαια δυσκολίες γιατί πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία, όπως ξέρετε, με ομοφωνία. Σε ό,τι αφορά την πρώτη πιτώρα ή την ενιαία διασάφηση ε, ή δήλωση, δεν συμφωνούμε. Μίλησε για ζήτημα επικουρικότητας ε, ο γερουσιαστής από τη Γαλλία. Η συνομική υπηρεσία όμως του Συμβουλίου είπε ότι δεν υπάρχει θέμα επικουρικότητας. Δεν ξέρω αν υπάρχει σχέση αιτίου αιτία του, αλλά όσο πιο πολύπλοκες γίνονται οι δηλώσεις ή διασαφήσεις, τόσο πιο μεγάλο ε, πρόβλημα έχουμε ε, απάτης ή μη ή ψευδούς δήλωσης, δηλαδή μεγαλύτερα έσοδα, αλλά δηλώνονται πολύ λιγότερα. Ο Δανός βουλευτής κύριος Γένσεν νομίζω μίλησε για την απλούστευση ή την απλότητα, αν θέλετε, του συστήματος. Στη Δανία που υπάρχει μόνο ε, ένας συντελεστής, ε, φορολογικός συντελεστής, 25% με μηδενικό συντελεστή για τις εφημερίδες. Εμείς θα το σκεφτούμε, θα το συζητήσουμε και με τα κράτη-μέλη. Και σας ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο, κυρία Πρόεδρε. Thank you very much. the panel... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα λοιπόν, ε, θα ήθελα να δεσολώσω τον κύριο Δεμετζόπουλο. Γιατί έχει και εκείνο να κάνει μια παρέμβαση. Ε, Πρόεδρε, ε, κυρίες και κύριοι, ο φόρο προστιθέμενη αξία αποτελεί μια από τι μεγαλύτερε πηγέ εσόδων για τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Λόγω όμω των διαφορετικών κανόνων που επικρατούν σε κάθε κράτο, η εισπραξή του καθώ και η επιχειρηματική δραστηριότητα σε διασυνοριακό επίπεδο καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο, μια και η συμμόρφωση αποτυγχάνει λόγω τη πολυπλοκότητα και του υψηλού κόστου τη διαδικασία οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια αποκλείει σαν επιλογή την αύξηση των συντελεστών άμεσης φορολογίας καθώς η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων έχει μειωθεί δραματικά. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα τη μεταβολή της φορολογικής επιβάρηση προς τους έμεσους φόρους όπως είναι και ο ΦΠΑ. Πολλά κράτη όπως και η Ελλάδα είχαν επιλέξει αυτήν την τακτική της αύξησης των έμεσων φόρων η οποία όμως προκάλεσε αύξηση στο τελικό κόστος των αγαθών και των υπηρεσιών και κατά συνέπεια μείωση στην κατανάλωση. Σύμφωνα με κάποια μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν δεν κάνω λάθος, το ύψος απώλειας των εσόδων από ΦΠΑ στην Ελλάδα αγγίζει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό για την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπερνάει τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η φορολογική λοιπόν της η μεταβολή της φορολογικής στρατηγικής προς έμεσους φόρους και η πολυπλοκότητα των διατάξεων που διέπουν το ΦΠΑ τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργούν φόρτο εργασίας επιχειρήσεις και εις δυσχέρειες στα κράτη-μέλη. Περισσότερο αυτό γίνεται αντιληπτό στις ενδοκινοτικές συναλλαγές όπου χρειάζεται να συντονίζονται τελείως διαφορετικά φορολογικά συστήματα. Η υιοθέτηση κοινών και σαφών κανονισμών που θα ενταχθούν στο νομικό καθεστώς των κρατών μελών θα βοηθούσε στην επίλυση των προαναφερομένων ζητημάτων. Όπως επίσης και θα μείωνε και το κόστος συμμόρφωσης στον ΦΠΑ. Μεταρρυθμίσεις σχετικά με την αναμόρφωση της δομής των φορολογικών συντελεστών την κατάργηση απαλλαγών λόγου χάρη για δημόσιους φορείς ή που αφορούν κοινωνικούς και πολιτιστικούς λόγους κρίνεται σκόπιμο να εξεταστούν ενδελεχώς αλλά και ο προορισμός του πεδίου εφαρμογής μειωμένων συντελεστών σε κοινά για όλα τα κράτη μέλη αγαθά και υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα κριτήρια. Η πρόταση οδηγία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υιοθέτηση τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ, την οποία επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών τη Ελλάδα, μπορεί να, να οδηγήσει στη μείωση του διοικητικού κόστου, στην ενίσχυση των δημόσιων ταμείων των κρατών μελών και στη διευκόλυνση της διασυνορικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και στην αναρμόνιση των κανόνων. Η πρόταση κατάργησης της δυνατότητας υποβολής ετήσιας δήλωσης ΦΠΑ χρησιμοποιείται ήδη από τη χώρα μου. Η Ελλάδα έχει εκφραστεί υπέρ της καταβολής του φόρου από τον προμηθευτή στον τόπο προορισμού όπω και υπέρ τη δημιουργία μηχανισμών ίσπραξη με τη μεσολάβηση των τραπεζών για την εξόφληση τιμολογίων και την άμεση καταβολή ΦΠΑ στο δημόσιο. Στο, σχέδιο, στο πεδίο των φορολογικών μεταρρυθμίσεων, η Ελλάδα έχει προχωρήσει στην απλοποίηση του φορολογικού κώδικα, υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων, κατάργηση του, κώδικα βιβλίων και στοιχείων, δημιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος διασύνδεσης των εφοριών, λογιστική έλεγχη βάση ανάλυση κινδύνου. Επειδή άκουσα και για το Eurofisk από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα συνεργάζεται με, την, ε, με το Eurofisk με όλες τις δυσκολίες που μπορεί να έχει όλο αυτό το είδους συνεργασία. Αυτό που έχει γίνει πάντως αντιληπτό είναι ότι υπάρχει έντονη ανάγκη αναμόρφωσης του υπάρχοντος συστήματος ΦΠΑ. Ένα σύστημα που ξεκίνησε το 1979 και πρέπει να αναμορφωθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να γίνει πιο απλοποιημένο και πιο αποτελεσματικό με ομοιομορφία διαδικασιών και κανόνων ανάμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα στη διαχείριση και διασταύρωση των πληροφοριών με στόχο την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής στις περιόδους αυτής της σοβαρής δημοσιονομικής στενότητας που διανύουμε η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής δεν είναι απλά ένα θέμα φορολογικής δικαιοσύνης αλλά αποκτά πια και ζωτική σημασία για την πολιτική και κοινωνική αποδοχή της δημοσιονομικής εξυγίασης από τους πολίτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, θυμάσαι που με ρώταγες αν καταλάβανα. Έχω μια άλλη κάρτα εδώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Θα ήθελα να σας μιλήσω για την Εστονία. Το σύστημα μας για το ΦΠΑ είναι τέτοιο με, που περιλαμβάνει ελάχιστες εξαιρέσεις και χρησιμοποιούμε το κλασικό επίπεδο. Μοιάζει με το δανέζικο σύστημα. Αλλά το κενό του ΦΠΑ υπάρχει και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Στην πράσινη βίβλο έχουμε διάφορα μοντέλα. για τη ε, νήσπραξη του ΦΠΑ και βασίστε στο γεγονός ότι προωθούνται οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Το λέω διότι η εστονική κυβέρνηση προβλέπει ένα μοντέλο όπου όταν το τιμολόγιο είναι ψηλότερο των χιλίων ευρώ οι πληροφορίες προωθούνται ηλεκτρονικά στις ε, φορολογικές αρχές. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι πόσο έχει προχωρήσει η Κομισιόν με τις μελέτες που αφορούν τα ζητήματα της πράσινης βίβλου σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των μοντέλων. Θα ήθελα να μάθω επίσης τι έχει επιτευχθεί σε σχέση με την πρόσβαση των κρατών μελών στα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στις βάσεις δεδομένων άλλων κρατών μελών. Το ρωτώ διότι η κυβέρνησή μας προσπαθεί να σχεδιάσει κάπως αυτό το μοντέλο και θα ήθελα να μου πείτε πόσο έχει προχωρήσει η Κομισιόν σε αυτές τις μελέτες και τι, πόσο αποτελεσματικές προβλέπετε να είναι. Πρόεδρος, έχουμε ακόμα δύο ομιλητές. Ε, ακούσαμε την Κομισιόν, δεν νομίζω θα επανέλθουμε για μια απάντηση. Ε, όλους φυσικά μας ενδιαφέρει αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών. Πιστεύω και η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. Θα θέλατε να επανέλθετε κύριε Βέρε, ότι είναι ένα θέμα που σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο. Δύο μικρέ παρατηρήσει θέλω να κάνω. Πρώτα απ' όλα να απαντήσω στα σχόλια της Κομισιόν. Μιλάτε για προβλήματα αρχής ε, όσον αφορά το σύστημα αντιστροφή τη επιβάρυνσης, το κατανοώ, αλλά δεν μπορούμε να προβλέψουμε το γεγονός ότι η αντιστροφή της επιβάρυνσης για το ΦΠΑ είναι ένα σωστό κατάλληλο πρακτικό εργαλείο που αναχαιτίζει τις απάτες ε, του ΦΠΑ ε, υπάρχει λοιπόν κάποια ε, πρόβλημα εδώ μεταξύ αρχής και πρακτικής. Ε, το δεύτερο, θα ήθελα να απαντήσω στο σχόλιο που κάνατε όταν αναφερθήκαμε στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών των εμπορευμάτων στην Ευρώπη. Για ορισμένα προϊόντα θα διατηρούμε πληροφορίες για την κυκλοφορία τους, για τη διακίνησή τους. Ε, σε γενικές γραμμές. Αν δείτε τα έσοδα από ΦΠΑ για ορισμένα προϊόντα, παρατηρείται απάτη στο ύψος του 10%. Δεν ζητάμε λοιπόν για συνεχείς τελωνιακούς ελέγχους ή παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας. Μιλάμε απλά για εχνηλασιμότητα των προϊόντων για να διατηρείται να διατηρούνται κάποιε πληροφορίε και κυκλοφορίε ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο παρατηρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μαρίνη. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ευχαριστήσω κυρίως τον πρόσωπο της Κομισιόν για τα στοιχεία που μας παρουσίασε πολύ συγκεκριμένα και να πω ότι και το θέμα που συζητούμε σήμερα είναι κατά μέρα το χαρακτηριστικό κλασικό θέμα όπου οι συζητήσει μεταξύ εθνικών βουλευτών και ευρωβουλευτών είναι χρήσιμο για να μην πω αναγκαίες, διότι βρισκόμαστε σε ένα τομέα κοινοτική νομοθεσίας, αλλά η εφαρμογή γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Και υπάρχουν πάρα πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, να αναλύσουμε, να διορθώσουμε. Επομένως, Επιθυμία μου θα ήταν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μετά τις σημερινές συζητήσεις να διατηρήσουμε τις επαφές μας για το θέμα του ΦΠΑ και την καταπολέμηση της απάτης, για τη βελτίωση της νομοθεσίας και για τις μεθόδους ελέγχου. Να συνεχιστεί λοιπόν η επαφή ε, και η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής σας αυτής, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τις ε, αρμόδιες εθνικές επιτροπές των κοινοβουλίων. Διότι νομίζω ότι πραγματικά με τον τρόπο αυτό αυτή η διακοινοβουλευτική διαδικασία μπορεί να λειτουργήσει και να συνεχίσει χωρίς να υπάρχουν προβλήματα σύγκρουσης αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκών, Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων. Φυσικά Είμαι διατεθειμένος να συζητήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος όλα αυτά τα θέματα, σε ό,τι αφορά την ενιαία δήλωση. Καταλαβαίνω ποιο είναι ο στόχος, ο στόχος είναι η απλούστευση, αλλά το να έχουμε μετάβαση από 26 σε 5 ε, παιδεία γιατί 26 είναι σήμερα στην Γαλλία, θα φτωχύνει κάπως, αν θέλετε, την πληροφόρηση και θα δώσει νέες, ε, θα ανοίξει νέα παραθυράκια για απάτη. Είναι όμως πειραματικό σας ακόμη αυτό, οπότε γιατί όχι, ας με πείσετε. Αν με πείσετε και δω ότι υπάρχουν ε, λογικά στοιχεία, μπορώ να το αποδεχθώ. Για να πω και στον Ολλανδανό συνάδελφο, κύριε Πρόεδρε, ότι το σύστημα αυτό με το μηδενικό συντελεστή και το συντελεστή του 25% κατ' εμέ είναι το βέλτιστο δυνατό. Είναι έτσι πολύ ισχυρό, σταθερό, πολύ καλό σύστημα κατ' εμέ για τα δημόσια οικονομικά. Στη χώρα μου υπάρχουν ε, κάποιες απόψεις ε, και προκαταλήψεις εγώ διαφωνώ. Θεωρώ ότι είναι καλό το σύστημα και μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε έτσι μεγαλύτερη ευελιξία και στην οικονομική ζωή, να συγκεντρώσουμε ε, τους πόρους μας και ιδανική εμπειρία για μένα είναι κάτι θετικό. Um, Σας ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς τώρα δεν έχουμε πια πάρα πολύ χρόνο. Βέβαια η συζήτηση ε, αποδείχθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Εάν τώρα η Επιτροπή επιθυμεί γραπτά να μας δώσει κάποιες απαντήσεις, ε, πολύ ευχαριστώ τις πληροφορίες αυτές μετά εμείς να τις διανύμουμε στα μέλη μας. Επειδή επιθυμούμε την περαιτέρω συνεργασία, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εξετάσουμε κυρίως ε, στην επόμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, θα ήταν λοιπόν ε, χρήσιμο να ε, συστήνουμε ομάδες εργασίας για συγκεκριμένα θέματα και πρέπει να πω ότι τελικά δεν είναι και αδύνατο να υπάρχει μια ομάδα εργασίας που να ασχολείται με τα φορολογικά και να συνεδριάζει ε, εξ αποστάσεως ε, με video conference, video διάσκεψη. Θεωρώ ότι κυρίως στην αρχή, οποτεδήποτε κανείς επιθυμεί την ανταλλαγή πληροφοριών, νομίζω επειδή τότε ακριβώ χρειάζεται κάνει πληροφορίε, αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Ε, και αυτό το καταθέτω ε, και ίσως ε, η γραμματεία μπορεί να το επιθυμήσει αυτό να το χρόνο στην επόμενη επιτροπή που θα σχηματιστεί με τη νέα θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι των εργασιών μας που είναι η δημοσιονομική εξυγίανση, η ανταλλαγή βέλτιστων δικών ε, και ξέρετε ότι πρόσφατα η έχουν εντοπιστεί οι προτεραιότητες ε, σχετικά με τη δημοσιονομική εξυγίανση για να προαχθεί η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα και για να εξυγχρονιστεί η δημόσια διοίκηση. Τα κράτη-μέλη ε, καλούνται να προβούν σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, να εξυγιάνουν τα δημόσια οικονομικά τους ε, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει κατανοητό με την έναρξη των νέων διαπραγματεύσεων το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μεγαλύτερη πολιτική υποστήριξη, το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της ε, μπορεί να προσφέρει καλύτερα κίνητρα για να προβούν τα μέλη, τα κράτη-μέλη ε, σε μεταρρυθμίσει. Επίσης αυτό που είναι σημαντικό είναι να γίνει κατανοητό ότι είδους μέθοδοι υπάρχουν έτσι ώστε να εντοπίζονται οι ε, περιτές δημόσιες ε, δαπάνες. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να υπάρξει καλύτερη εξυγίανση των δημοσιονομικών και να εφαρμοστούν βέλτιστες πρακτικές στα κράτη-μέλη. Θεωρώ λοιπόν ότι μάλλον ε, εδώ θα έχουμε κάποιους ομιλητές εδώ στο πόντιουμ. Δύο-τρία λεπτά να κάνουμε διάλειμμα για να ξανα τα βρούμε εδώ πάνω στο μου να έρθουν αυτοί που πρέπει να έρθουν. Αν έχετε καλοσύνη, ε, στείλτε μας ε, όσο δυνατόν ε, συντομότερα τις ερωτήσεις σας. Υπάρχουν διάφορες κάρτες που κυκλοφορούν, άσπρες ή ροζ, και εμείς θα σας δώσουμε το λόγο. Σε δύο-τρία λεπτά επανερχόμεθα. Ωραία λοιπόν, να συνεχίσουμε με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και υπάρχει καφές έξω για όσους το επιθυμούν. Καλωσορίζω τους ομιλητές, ε, η κυρία Κόραν Εβενχάουζεν, είμαι σίγουρο ότι το σκότωσα το όνομα, από το Ολλανδικό Κοινοβούλιο και ο κύριος Βιντσέντι Μαρτίνες Πιάντε από το από την Ισπανική Βουλή και θα μας περιγράψουν τις δικές τους απόψεις και τις δικές τους εμπειρίες. Έχετε το λόγο, Κόρα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Μετά από πενταετές διάστημα αρνητικής ή ε, ελληματικής ανάπτυξης φαίνεται να αναστρέφεται η τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι στατιστικές υπηρεσίες δείχνουν ε, στοιχεία ανάκαμψης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να τροφοδοτήσουμε ως κράτη-μέλη αυτή την ε, ανάπτυξη εξηγένοντας τους προπολογισμούς και τις οικονομίες. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν τις ιδιαιτερότητές τους, τα δικά τους χαρακτηριστικά και τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, συνεπώ χρειάζεται λύσεις προσαρμοσμένες στο εκάστοτε κράτος μέλος. Δεν υπάρχει μία λύση ενιαία για όλους. Οι Ολλανδοί πολίτες αισθάνονται επίσης τις επιπτώσεις της οικονομική κρίσης. Οι ανεργίε στις κατοχώρε είναι υψηλή για τα δικά μας δεδομένα. Επιπροσθέτως, οι κατοχώρε ε, έχουν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της γύρασης του πληθυσμού που μπορεί να δημιουργήσει μακροπρόθεσμα προβλήματα εάν δεν εφαρμοστούν μεταρρυθμίσεις μεταξύ άλλων και στο σύστημα υγεία μα. Οι κάτω έχουν επίση να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των υψηλών τιμών ε, των ακινήτων ε, και τη συμφόρηση τη αγορά ακινήτων. Και ε, παρατηρείται και αύξηση των δαπανών σε και Χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσει για καλύτερη παροχή των κοινωνικών μας παροχών. Οι μεταρρυθμίσεις επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών. Είναι καθήκον λοιπόν εμά, των πολιτικών να εξηγούμε στου πολίτε για ποιο λόγο αυτές οι σκληρές μεταρρυθμίσεις του συμφέρουν. Η σημαντική πρόκληση είναι να έχουμε την υποστήριξη των πολιτών για αυτές τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Να μοιραστώ μαζί σας δύο σημαντικές βέλτιστες πρακτικές ε, που έχουμε στις ε, κατοχώρες, στις ευρείες ε, συμφωνίες και την αποκέντρωση Πρόσφατα στις κατοχώρες ε, συνέχισαμε συμφωνίες μεταξύ κυβέρνησης, ε, κοινοβουλίου, εργοδοτών, εργαζομένων και κοινωνιών των πολιτών. Ε, αφορούν μεταρρυθμίσεις στις συντάξει, στις κοινωνικές υπηρεσίες, στη στέγαση και την υγειονομική περίθαλψη. Προσπαθήσαμε να βρούμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ της ευρείας υποστήριξης των μεταρρυθμίσεων, του ρυθμού των μεταρρυθμίσεων και τη οικονομική σταθερότητα. Δεύτερον, επιλέξαμε όπου ήταν δυνατόν να εκτελούνται οι μεταρρυθμίσεις στο χαμηλότερο δυνατό δημόσιο επίπεδο, δηλαδή κοντά στους επηρεαζόμενους πολίτες. Για παράδειγμα, η, εκτέλεση, η υλοποίηση του νέου συστήματος φροντίδας για τους νέους ε, ε, έχει αποκεντρωθεί σε επίπεδο δήμων. Έτσι διασφαλίζεται ότι όσον αφορά την ανάπτυξη των παιδιών μας, παράγοντες όπως το οικογενειακό περιβάλλον, η εκπαιδεία, η ασφάλεια και τα αθλήματα λαμβάνονται ακόμη καλύτερα υπόψη. Οι Δήμοι επίσης ε, αναλαμβάνουν την ευθύνη της εφαρμογής των μακροπρόθεσμων πολιτικών φροντίδας μας διότι αυτοί μπορούν καλύτερα να κρίνουν κατά πόσο είναι απαραίτητη η φροντίδα που ζητείται κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να συνεχίσω με κάποιε παρατηρήσει για το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω μεσοτόνωση των μεταρρυθμίσεων. Η εσωτερική αγορά βρίσκεται στην καρδιά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει παρουσιάσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τι κατοχώρε, διότι πολλέ από τι θέσει εργασία μα εξαρτώνται από αυτό. Καλέ εποχέ για την Ευρώπη σημαίνει καλέ εποχέ για τι κατοχώρε. Από την άλλη, όμω, η οικονομική κρίση στην Ευρώπη γίνεται άμεσα αισθητή στι κατοχώρε. Έτσι λοιπόν ε, η πλειοψηφία του Ολλανδικού Κοινοβουλίου θεωρεί απαραίτητη την οικονομική σύγκληση. Παρ' όλα αυτά το Ολλανδικό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων παραμένει εθνική αρμοδιότητα. Τα επιμέρους κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να κάνουν τις δικές τους επιλογές πολιτικής έχοντας στο νου τους ότι αυτές τους συμφέρουν. Πριν από το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ολλανδικό Κοινοβούλιο συζήτησε σε βάθος την ενίσχυση του συντονισμού πολιτικών. Έγινε μια συζήτηση όσον αφορά τις ε, συμβατικές διευθετήσεις και τις δυνατότητες μηχανισμών αλληλεγγύης. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ολλανδικό Κοινοβούλιο έκανε έκκληση στην κυβέρνηση να απορρίψει την εισαγωγή νομικώς δεσμευτικών ε, συμβατικών διευθετήσεων, στο ε, πλαίσιο των πολιτικών μέτρων και των μεταρρυθμίσεων. Όσον αφορά τους μηχανισμούς αλληλεγγύης, υποστηρίζουμε τους προσανατολισμούς στους οποίους συμφώνησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θεωρούμε ότι οι μηχανισμοί δεν πρέπει να συνεπάγονται υποχρεώσεις για κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν στο σύστημα αμοιβαία συμφωνημένων συμβατικών διευθετήσεων. Δεν πρέπει να γίνουν εργαλείο εξίσωση των εσόδων, ούτε να επηρεάσουν το πολιτισμικό πλαίσιο. Θα πρέπει να ε, σέβονται την ε, δημοσιονομική κυριαρχία των κρατών μελών. Αναμένουμε την περαιτέρω εμβάθυνση και τις ιδέες του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επί του θέματος και σίγουρα θα συνεχίσουμε με κάποιες ε, σε βάθος συζητήσεις γι' αυτό. Δεδομένου του περιορισμένου χρόνου, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και προσβλέπω στις συζητήσεις μας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Περνάω τώρα στον κύριο Βιντσέντε Μαρτίνες από το Ισπανικό Κογκρέσο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να παρέμβω σε αυτή την ε, συνέλευση και θα ήθελα να σας παρουσιάσω τις δικές μου σκέψεις από την επιτυχή εμπειρία που είχαμε εμείς στην Ισπανία τα τελευταία δύο χρόνια. Η, κατά την άποψή μου, ο συντονισμός ε, και η ομογενοποίηση των οικονομικών πολιτικών των χωρών της Ένωσης είναι βασικό, βασική προϋπόθεση για να έχουμε μια οικονομική συνοχή που θα επιτρέπει τη διατήρηση και τη σταθερότητα του ευρώ. Με την κρίση ε, καταδείχθηκε ότι δεν είναι αμετάκλητο το ευρώ και για να διατηρηθεί θα πρέπει να υπάρχει οικονομική ισορροπία σε κάθε μια από τις χώρες μέλη. Είναι πολύ σημαντική η οικονομική πολιτική που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αλλά ταυτόχρονα είναι αναγκαίος ένας μεγαλύτερος συντονισμός των πολιτικών ε, κάθε μιας από τις χώρες μέλη, ώστε να έχουμε μια βιώσιμη ε, οικονομική ανάπτυξη με συνοχή. Και η δουλειά που γίνεται στις εμμονωμένες χώρες επηρεάζει και το σύνολο. Δηλαδή, αυτή η Επιτροπή για την Οικονομική Διακυβέρνηση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Από τότε που ξέσπασε η κρίση και τα κρατημέλη αλλά και οι χώρες Ευρωζώνης έλαβαν διάφορα μέτρα και κατέληξαν σε συμφωνίες για την εφαρμογή και την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής και για την αποτροπή μιας παρόμοιας κρίσης στο μέλλον. Όμως, πρέπει να υπάρξει συντονισμός των οικονομικών πολιτικών, να υπάρξει μια ενιαία εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να εφαρμοστούν παρόμοιε απαιτήσει ε, στι ε, χρηματοοικονομικές ε, οντότητε και στι επιχειρήσει όλων των χωρών. Στις 13 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την ετήσια προοπτική μελέτη για την ανάπτυξη και έτσι δρομολογήθηκε επισήμω και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο του 2014. Σε αυτή λοιπόν την ετήσια επισκόπηση ε, ανάπτυξη αναφέρονται πέντε βασικέ προτεραιότητε. Ο δρόμο είναι σωστό, αλλά πρέπει να τον προχωρήσουμε. Να τον διαβούμε. Στην Ισπανία η κρίση που ξέσπασε για πρώτη φορά το 2007 επειδή είχαμε επεκτατικέ πολιτικέ ε, σε ό,τι αφορά τι δημόσιε απάνε, ενώ δεν υπήρχαν και διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει για βελτίωση τη ανταγωνιστικότητα, όλα αυτά οδήγησαν ε, στα όρια τη στην Ισπανία. 12% το εξωτερικό έλλειμμα, δημόσιο έλλειμμα που είχε φτάσει κάποια στιγμή το 10% και διαρθρωτικά παγιώθηκε γύρω στο 7% και με ποσοστά ανεργίας πάνω από το 25%. Οι δυσκολίες των αγορών και η κρίση χρέους έκαναν ανέφικτη τη χρηματοδότηση της οικονομίας και τα επιτόκια κινδύνου ανέβηκαν σε τεράστιες, σε δυστεώρητα ύψη. Και έτσι χρειάστηκε να εφαρμόσουμε ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα προσαρμογής μετά από τις ε, ε, εκλογές ε, τον Νοεμβρίου 2011 με πολύ μεγάλη πλειοψηφία εξελέγει στην κυβέρνηση το Λαϊκό Κόμμα. Προσαρμογή λοιπόν για την μείωση, ε, τη σταθερή μείωση του δημόσιου χρέους και ελλείμματος και βέβαια τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω μεταρρυθμίσεων. Κατά την άποψή μου, οι μεταρρυθμίσεις πραγματικά μεταμόρφωσαν ε, την αγορά εργασία, το εκπαιδευτικό σύστημα, τη δημόσια διοίκηση, τι αγορέ αγαθών και υπηρεσιών στην Ισπανία. Ενίσχυσαν και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η Ισπανία έτσι μπόρεσε να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της, να βελτιώσει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία της και να πάψει να είναι ένα πρόβλημα για τη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Επίσης, οι αναπτυξιακές προοπτικές για το 2014 βελτιώθηκαν θεαματικά, όπως το είδαμε και το ακούσαμε χθε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αφήσαμε πίσω μας λοιπόν ως χώρα την ύφεση. Το τελευταίο τρίμηνο είχαμε αύξηση στα τριμηνία στοιχεία 0,7%. Το 2013 μειώθηκε η ανεργία κατά 147.385 άτομα. Τα ασφάλιστρα κινδύνου είναι κάτω από τα 200 από τους 200 πόντους, αυτό δεν το είχαμε δει από το Μάιο του 2011 και μετά, οι ξένες επενδύσεις σχεδόν διπλασιάστηκαν και οι εξαγωγές δείχνουν ένα πολύ μεγάλο δυναμισμό. Έχουμε αύξηση δάξεως με την εμπειρία μας αυτή λοιπόν θεωρούμε ότι στις χώρες Ευρωζώνης πρέπει να γίνουν περισσότερες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, αλλά όλες πρέπει να βαθίζουν προς την ίδια κατεύθυνση. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ απαιτητικοί με τη δημοσιονομική εξυγίανση και με την υποχρέωση να διατηρήσουμε τα δημόσια ελλείμματα γύρω στο 3%. Και επίσης θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε σκέψεις όπως ότι με το ευρώ είναι εγγυημένη, ισορροπημένη ανάπτυξη ή ότι μπορούν να είναι τα επιτόκια παρόμοια σε όλες τις χώρες. Διότι αυτό αποδείχθηκε ότι δεν είναι βέβαιο. Ναι. Και στην Ισπανία εμείς καταλάβαμε ότι η κρίση μπορεί να είναι χρήσιμη υπό την έννοια ότι μπορεί να μας κάνει να είμαστε πιο απαιτητικοί σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των οικονομικών πολιτικών και την υλοποίηση πιο εντατικών μεταρρυθμίσεων. Εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να πιστέψω ότι η Ευρώπη είναι μια οικονομική ζώνη που δεν έχει μέλλον. Πιστεύω ότι αν τα καταφέρουμε έχουμε τεράστιο, τεράστια δυναμική όλες οι χώρες μαζί και το κράτος πρόνοιας είναι ένα στοιχείο συνοχής που καθιστά βιώσιμη αηφόρο την ανάπτυξη. Η άποψή μας στην Ισπανία και η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι αν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί προχωρήσουμε μαζί και στη σωστή κατεύθυνση θα αναπτυχθούμε από κοινού και θα είμαστε από τις πλέον ανταγωνιστικές και με τις μεγαλύτερες δυνατότητε περιοχές του δυτικού κόσμου. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον κύριο Αλέξανδρο Μετζόπουλο ξανά. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, πάνε σχεδόν έξι χρόνια από το ξέσπασμα τη διεθνού χρηματοπιστωτική κρίση και η οικονομική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακόμα εύθραυστη οι οικονομίε ορισμένων χωρών χαρακτηρίζονται από ύφεση, ενώ το ποστό ανεργία στη ζώνη του ευρώ ξεπερνάει το 11%, με την ανεργία των νέων σε κάποιε χώρε να αγγίζει σε μη βιώσιμα πια επίπεδα. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένα χάσμα ανταγωνιστικότητα ανάμεσα στι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο, η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική επιτάχυνση στη δημοσιονομική εξυγίανση βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε διάφορους τομείς. Η δημοσιονομική προσαρμογή που έχει πετύχει η χώρα μου μεταξύ του 2009 και του 2013 είναι η πιο γρήγορη και μεγαλύτερη που έχει πετύχει ποτέ χώρα του ΩΣΑ με μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης κατά 13,4 ποσοστιαίες μονάδες επί του ΑΕΠ, μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος κατά 10,8 μονάδες, το πρωτογενές πλεόνασμα, κύριε και κύριοι βουλευτές, στο τέλος του 2013 εκτιμάται στο 0,4% ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει διαρθρωτικό πλεόνασμα 1,2% του ΕΕ για το ίδιο διάστημα. Συνολικά, τα δύο τρίτα της απαιτούμενης δημοσιονομικής προσαρμογής για τη μείωση του χρέους σε βιώσιμα επίπεδα ως το 2020 έχει ήδη επιτευχθεί με τα μέτρα να μοιράζουν ισότιμα ανάμεσα σε περικοπές δαπανών και σε αυξήσει φόρων. Αναφορικά με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ενδεικτικά μόνο θα σας αναφέρω ότι έχει γίνει μεταρρύθμιση στο συνταξιδοτικό σύστημα με μείωση της μέσης σύνταξης αλλά κυρίως των ψηλών συντάξεων κατά 40%, αύξηση του ορίου ηλικία συνταξιοδότησης και απαιτούμενων συνολικών ετών εργασίας στον τομέα της αγοράς εργασίας έχει καθοριστεί νέος μηχανισμός κατώτατου μισθού, ε, ρύθμισης κατώτατου μισθού περικοπές μισθών στο δημόσιο τομέα και μείωση του χρόνου ζωής των συλλογικών συμβάσεων. Στη δημόσια διοίκηση, η μεταρρύθμιση προχώρησε με μείωση των απασχολούμενων, με ενιαίο μισθολόγηση και με διαρκή αξιολόγηση των υπαλλήλων. Έχουμε μεταρρυθμίσει την τομέα υγεία με συγχώνευση των οκτώ υπαρχόντων ασφαλιστικών φορέων και ταμείων σε ένα, που καλύπτει πια σχεδόν όλο τον πληθυσμό, με έλεγχο τη επίδοση των νοσοκομειακών μονάδων, με ευρύτερη χρήση των γενώσιμων φαρμάκων και με εισαγωγή ενό συστήματο ηλεκτρονική συνταγογράφησης. Έχουμε μεταρρυθμίσει στην νομία τη κοινωνική προστασία που περιλαμβάνουν τον εξορθολογισμό των κοινωνικών επιδομάτων και τον σχεδιασμό πολιτικών για τους μακροχρόνιου άνεργου. Ε, στο δημοσιονομικό τομέα ακόμα περιλαμβάνεται ενισχυμένο δημοσιονομικό πλαίσιο για έλεγχο και αυτόματο μηχανισμό διόρθωσης όταν δεν πάνε καλά τα οικονομικά. Τέλος, ο κατάλογος που δεν τελειώνει των μεταρρυθμίσεων που έχουν γίνει στη χώρα μου τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει την απελευθέρωση των οδικών μεταφορών, το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων και μια σειρά από άλλα τέτοια μέτρα. Όλα αυτά όμως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχουν μια τρομακτική συνέπεια. Η συνέπεια αυτών των μεταρρυθμίσεων τα τελευταία χρόνια, όπου ο ΩΣΑ καθορίζει και κατατάσσει την Ελλάδα σαν μια από τις πιο φιλικά χώρες ε, προς την ανάπτυξη έχουν μια τρομακτική συνέπεια. Το 2013 ήταν η έκτη συνεχόμενη χρονιά ύφεση για τη χώρα μου με δραματική μείωση του ΑΕΠ πάνω από 25% με δραματική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικοκυριών πάνω από 40% με αλματώδη αύξηση ανεργίας πάνω από 27% και σε ορισμένε περιπτώσεις πάνω από 60% για τους νέους. Με μείωση της βάσης των καταθέσεων, πράγμα που περιορίζει την παροχή ρευστότητα ακόμα και προσεγγίσεις υγιεί επιχειρήσεις. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, όσον αφορά το θέμα που συζητάμε, συγκεκριμένη συνταγή για κατάλληλο μείγμα ανάμεσα στη δημοσιονομική εξυγίανση και πολιτικές που προωθούν την ανάπτυξη δεν υπάρχει. Εξαρτάται από τη διαφορετική δημοσιονομική και οικονομική κατάσταση κάθε χώρας καθώς και το ρυθμό προσαρμογής της στην προσπάθεια οικονομικής σταθεροποίησης και στην εφαρμογή διαρθρωτικών πολιτικών. Κρίνεται όμως απαραίτητο στη λήψη όλων αυτών των σχετικών αποφάσεων η κάθε χώρα να αξιολογεί το μέγεθος της αναγκαίας δημοσιονομικής λιτότητας, τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο σύνολο της οικονομίας, τις κοινωνικές ανισότητες και την κοινωνική συνοχή, τις υποδομές και τη διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα και τέλος τις συνθήκες χρηματοδότησης της δική τη οικονομίας. Κυρίως όμως αυτό το οποίο θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη είναι τα δικά της χαρακτηριστικά. Κάθε χώρα έχει το δικό της DNA, κάτι το οποίο δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η ευρωπαϊκή ένωση μέσα από τις πολιτικές της μπορεί να συνεισφέρει καταλυτικά στις προσπάθειες κάθε κράτους μέλους για την επιστροφή τους στην ανάπτυξη και για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. δράσεις όπως είναι η μείωση του βασικού επιτοκίου σε χαμηλά ε, επίπεδα από την ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα ενίσχυση των μικρομεσαίων με χρήση ε, μέρους από του πόρου των διαρθρωτικών ταμείων ω εγγυήσει για νέα τραπεζικά δάνεια και ακόμα η χορήγηση δανείων σε κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που αντιμετωπίζουν δυσκολίε και εφαρμόζουν σκληρέ δημοσιονομικέ πολιτικέ είναι μέτρα σε μια σωστή κατεύθυνση. Η επιστροφή στην ανάπτυξη, ιδίω για τα κράτη-μέλη που αντιμετώπισαν χρόνια ύφεση, όπω και η δημιουργία θέσεων εργασία και η βελτίωση των συνδικών ρευστότητα, είναι υψίστη σημασία για ευνόητου οικονομικού αλλά και κοινωνικού, κρατικού και λόγου σταθερότητα πρέπει να αποτελούν πλέον βασική προτεραιότητα των πολιτικών που χαράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό, ανεξάρτητα από τι συνθήκε που βιώνει κάθε κοινωνία, οι πολιτικέ προσαρμογής που εφαρμόζονται να είναι προσανατολισμένε στην ενίσχυση τη κοινωνική συνοχή, να συνδυάζονται με αναπτυξιακέ πολιτικέ και φυσικά να εντάσσονται στι κατευθύνσει τη στρατηγική Ευρώπη 2020, καθώ και στι βασικέ αρχέ τη ίδρυση αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. Προσπαθώ να παροτρύνω και άλλους να στείλουν το χαρτάκι τους για να μπορούν θέλουν να μιλήσουν. Πρώτα απ' όλα λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο Θεοδόρ Στοιν ο οποίος είναι ιδιαίτερα δραστήριος ε, σε πολλά ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ ήμουν υπουργό οικονομικών, υπήρξα υπουργό οικονομικών στη Ρουμανία. Εκείνη την εποχή διαπραγματεύτηκα πολλέ ε, συμφωνίε για την αναδιάρθρωση τη ρουμανική οικονομία με το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο εκείνη την εποχή. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι προηγουμένως. Η κάθε χώρα είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Παρ' όλα αυτά οι πολιτικοί δεν φαίνεται να κατανοούν ότι όταν ε, έχει κάποιος να αντιμετωπίσει προβλήματα στην οικονομία της χώρας του ε, έχει χάσει ανταγωνιστικότητα, έχει υπερβολικά υψηλό χρέο και χρειάζεται προσαρμογή. Η προσαρμογή αυτή είναι πόδινη. Ναι. Αυτή η διαδικασία ε, προσαρμογής ε, δεν έχει κάποια αναλλακτική λύση. Αυτό που κάναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο επίπεδο των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων ήταν ότι εκφράσαμε αλληλεγγύη που επικουρείται όμως και από ευθύνη, από ανάληψη ευθύνης, διότι το πρόβλημα οποιοδήποτε προγράμματος προσαρμογής είναι ότι πρέπει να δώσει στη χώρα τον χρόνο που χρειάζεται για να εφαρμόσει τα μέτρα αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητάς της. και οι πιστωτέ ε, θα πρέπει να παρέχουν στην εκάστοτε χώρα τον απαραίτητο χρόνο ώστε να μπορέσει να εξισορροπήσει αφενός τις ε, δεσμεύσεις πληρωμών και από την άλλη τις πραγματικές δυνατότητες ε, καταβολής πληρωμών. Δυστυχώς η διαδικασία αυτή που χρειάστηκε αρκετά χρόνια υπήρχε κάτι το οποίο δεν λειτουργήσε ακριβώς όπως προβλεπόταν δεν ε, είχαμε αξιολογήσει σωστά τις δυνατότητες ε, πληρωμής της ε, συγκεκριμένης χώρας και τις απαιτήσει αναδιάρθρωσης των πληρωμών. Και φυσικά μερικές φορές χρειάστηκε στην πορεία της να προσαρμοστεί, να διορθωθεί αυτή η διαδικασία και χρειάστηκε να προσθεθούν νέοι πόροι. Θα έχετε παρατηρήσει ότι όλη η συζήτηση που είχε γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή την έκθεση ε, που αφορά το ρόλο που διαδραμάτισε η Τρόικα και τα προβλήματα σεβασμού της κυριαρχίας και της δημοκρατίας ε, θα τα έχετε παρατηρήσει. Ε, καλό είναι που τα συζητάμε όλα αυτά, κατά την απόψή μου. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι μια χώρα που δεν μπορεί να συνάψει δάνεια με εύλογους, χώρους, με εύλογους όρους χρειάζεται να προσαρμοστεί. Ευχαριστώ Πρόεδρος. Από το Ισπανικό Κογκρέσο έχουμε τον Πέντρο Σάουρο. Ah, Σας ευχαριστώ. Σύντομα. Αυτό που με ανησυχεί τα μάλα Είτε ότι μιλάμε για την απονοποίηση, αν θέλετε, της ε, ευρωπαϊκής οικονομίας. Και θεωρώ ε, ότι οι διαθροτικές μεταρρυθμίσεις θα έπρεπε να είναι συμβατές με τον οικονομικό κύκλο της κάθε χώρας και συμβατές με την δημοσιονομική εξυγένση. Και σας δίνω ένα παράδειγμα. Εάν γίνει μια μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, όπως έγινε στη χώρα μου, που συνεπάγεται πιο φτηνές απολύσεις και μικρότερους, χαμηλότερους μισθούς. Αυτό περιπλέκει τη δημοσιονομική εξυγίανση. Γι' αυτό και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ε, και αυτή τη, αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή Όλες ε, οι πολιτικές μπορεί να έχουν ως στόχο την έξοδο από την κρίση, αλλά κάποια μέτρα μπορεί, όπως είπα, να περιπλέξουν τη δημοσιονομική εξηγένση. Πρέπει λοιπόν να βρούμε και την κατάλληλη χρονική στιγμή για καθένα από τα μέτρα. Αυτό είναι μια σημαντική ιδέα. Δεν είναι δική μου βέβαια. Υπάρχει ένα σημαντικό ρεύμα, μια σχολή σκέψης. Το Δούνου για παράδειγμα, δίνει έμφαση σε αυτές τις συνθήκες καλές πρακτικές για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν οι κατάλληλες και αποτελεσματικές πολιτικές που θα φέρουν αποτελέσματα. Δεύτερον, δεύτερη ιδέα, δημοσιονομική εξηγένση. Θα ήθελα να ακούσω να γίνεται περισσότερο λόγος για μεσοπρόθεσμα προγράμματα δημοσιονομικής εξηγένσης που θα είναι αξιόπιστα και θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα, όχι μόνο στο σκέλος των δαπανών, αλλά και στο σκέλος των εσόδων. Και όπως είπα πρέπει να αξιολογούνται τα προγράμματα αυτά από ανεξάρτητες, πραγματικά ανεξάρτητες αρχές που να μην έχουν καμία σχέση με τις κυβερνήσεις. Να εξαρτώνται αν θέλετε περισσότερο από τα κοινοβούλια και όχι τόσο από τις κυβερνήσεις στη χώρα μου. Η διοίκηση αυτή εξαρτάται περισσότερο από την κυβέρνηση και όχι τόσο από το κοινοβούλιο. Παραλαμβάνω, αξιόπιστη πρέπει να είναι η δημοσιονομική εξυγένση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για το προηγούμενο έτος, το 2013, θα σας δώσω δύο στοιχεία. Η κυβέρνηση είχε θέσει στόχους για το έλλειμμα 3,8 για το 2013. Όμως το Σεπτέμβριο του 2013 σε με του Σεπτέμβριο του 2012, λαμβάνοντας υπόψη τις ε, ενισχύσεις τις οικονομικές, 10,3 ήταν το έλλειμμα. Και το χρέος, άλλο στοιχείο, που το έχω σχολιάσει ξανά, το δημόσιο χρέος σε δύο χρόνια αυξήθηκε κατά 23%. Και άλλα 30, άλλες 30 ποσοστίες θα ανεβεί τα επόμενα χρόνια. Επομένως, θα ανέβει τα 30. Δηλαδή, ε, πραγματικά, η στιγμή αυτή είναι ιστορική. Πρέπει και μπορεί να αλλάξει η Ευρώπη. Αλλά πρέπει να κάνουμε καλά τα πράγματα και με διαφορετικό τρόπο για να μπορέσει η Ευρώπη να βγει με πιο στεναρό τρόπο, πιο δυνατή από την κρίση, να δημιουργήσει αλληλεγγύη, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Από την Ολλανδική Γερουσία, ε, Ρενέ Βαντελίντεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. στα, τρία, στα κράτη-μέλη συχνά η συμμετοχή του το 3% προέρχεται από τις Βρυξέλλες ενώ προέρχεται από τα ίδια τα κράτη-μέλη διότι τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που όρισαν ότι η υλοποίηση του 3% για τους ε, ε, πολίτες, ε, για τις θέσεις εργασίας, για τη σταθερότητα και για την ανταγωνιστικά των κρατών μελών στο μέλλον είναι η καλύτερη προσέγγιση. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν Μην δίνουμε δηλαδή στους πολίτες ε, την εντύπωση ότι μιλάμε για παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας όταν οι ίδιοι ε, όρισαν ε, κάτι τέτοιο. Επιβάλλουμε υποχρεώσεις. Αληθεύει. Σημαίνει ότι έχουν λιγότερο περιθώριο λεγμών τα κράτη-μέλη. Πρέπει τα κράτη-μέλη να κάνουν ε, τις επιλογές τους εντός αυτού του ορίου του 3%. Το κατά πόσο συζητάμε για νομική πολιτικά δεσμευτικές υποθέσεις όχι. αυτή είναι μια πολιτική δέσμευση. Ε, στο μέλλον Κάποια κράτη-μέλη μπορεί να το κάνουν γιατί συμβαίνει θα το κάνουν εις βαρος άλλων κρατών μελών. Τα εθνικά κοινοβούλια λοιπόν πρέπει να συνεργαστούν με τα υπόλοιπα ε, κοινοβούλια και πρέπει να τηρούν τις δεσμεύσεις τους στα κράτη-μέλη. Και όταν μιλάμε για κυριαρχία, αυτή η συζήτηση έχει γίνει πολύ συχνά στα κράτη-μέλη για τους λάθους λόγους. Πρέπει να δούμε τι εννοούμε με τον όρο κυριαρχία. Κυριαρχία τι σημαίνει ότι ε, αναλαμβάνει κάποιο την ευθύνη των δικών του υποθέσεων. Ε, οι πολίτες βλέπουν ότι λαμβάνουμε μια απόφαση και ότι αυτή επηρεάζει όσοι συζητάμε. Σε διάφορους τομείς ε, αυτό έχει τελειώσει. Όταν μιλάμε για εμπόριο, για την εμπορική πολιτική, για παράδειγμα, για την νομισματική πολιτική, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μην δίνουμε την ευκαιρία στους λαϊκιστές να λένε ότι θέλουν να καλύπτουν την πραγματικότητα. Διότι αυτό που είναι καλύτερο για την Ευρώπη είναι καλύτερο και για τους πολίτες της Ευρώπης, της κάθε χώρας και για το μέλλον εντός των ορίων που υπάρχουν έχουμε κάποιο περιθώριο ελιγμών ε, εθνικά πιο περιορισμένο. Πρέπει να φροντίσουμε να διασφαλίσουμε ότι όταν μιλάμε για σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας να μην ε, δημιουργούμε την εντύπωση ότι είμαστε κύριοι των δικών μας υποθέσεων. Είμαστε συνδεδεμένοι ο ένας με τον άλλο και αλληλοεξαρτώμενοι μέτρα που λαμβάνονται σε ένα κράτος μέλος έχουν συνέπειε σε ένα άλλο κράτος μέλος. Καλό είναι λοιπόν που αυτή τη βδομάδα έχουμε εδώ βουλευτές από όλες τις χώρες που συναντώνται και φροντίσουμε να συνεννοηθούμε, να πούμε ότι πρέπει να ε, μοιραστούμε τις ευθύνες ε, για τις πολιτικές, για τις μελλοντικές πολιτικές των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ε, thank you Σας ευχαριστώ πολύ. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Αντολίν Σάντσεφ Πρεσέδο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να κάνω μια παρέμβαση για τις βέλτιστες πρακτικές και να χαιρετήσω την παρέμβαση του συμπατριώτη μου, ο οποίος μίλησε για την κατάσταση στην Ισπανία, ο Βιθέντε Μαρτίνιθ που χάλεται συγκεκριμένα. Πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση σε κάποιες πτυχές όμως που δεν ε, τονίστηκαν επαρκώς. Πρώτον, ότι τα κράτη-μέλη είναι σε καλύτερη θέση να δώσουν απαντήσεις στις τεράστιες προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν. Πρώτον, όταν υπάρχουν σημαντικές εσωτερικές συμφωνίες, όταν έχουν δεσμευτεί οι βασικές πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Και δεν θα πρέπει ε, να μιλάμε με μεροληπτικό τρόπο και μη αντικειμενικό για τη γένεση της κρίσης και την αντιμετώπιση της. Όλοι μας ξέρουμε θα μπορούσε να έχει αποτραπεί με μια νομισματική, με μια δημοσιονομική πολιτική πιο αυστήρη. Επομένως ε, πρέπει να ε, αφήσουμε κατά μέρο όλα όσα ακούγονται από διαφόρους. Θέλω να τονίσω ότι η Ισπανία είναι μια χώρα η οποία πράγματι, πράγματι είχε εφαρμόσει επεκτατικές πολιτικές ε, ως απάντηση στο πρώτο κύμα της κρίσης, αλλά το έκανε ε, σε ένα πλαίσιο ε, εκκλήσεων από πλευράς G20. Και επειδή υπήρχαν κράτη-μέλη που είχαν μια κατάσταση δημοσιονομική που είχαν τη δυνατότητα να, κάνουν μια όθηση, το, να έχουν μια όθηση, το έκαναν. Και εκεί το πρόβλημα της διεθνούς δέσμευσης ε, τίθεται και είναι πάρα πολύ σημαντικό για να διατηρηθεί η οικονομία μέσα στην οποία κινούμαστε και εμείς. Νομίζω ότι είναι σημαντικό ε, στο ευρωπαϊκό επίπεδο να αξιολογήσουμε και να βάλουμε στο σωστό ε, πρίσμα αυτά τα οποία έγιναν τους τελευταίους μήνες υπήρχε μια αυτοπροκαλούμενη θα έλεγα ύφεση λόγω των λανθασμένων πολιτικών. Υπήρχαν κάποια σμεροληψίες, κάποια συστηματικά ε, σφάλματα ε, Πάντως καταφέραμε να ξεπεράσουμε την ύφεση με πιο μετριοπαθή στοιχεία πλέον και τώρα καταφέρνουμε από το 2011 και μετά να βγούμε από το τέλμα. Και είναι η δεύτερη τόσο δύσκολη κρίση που ξεπερνάμε μετά το τέλος του εμφύλιου πολέμου. Υπάρχουν στόχοι του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, τις μακροοικονομικές ανισορροπίες είναι και οι στόχοι της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020 που πρέπει να επιτύχουμε. Δεν πρέπει όμως ε, να ε, πούμε ότι έχουμε θριαμβεύσει. Αντίθετα πρέπει να είμαστε πολύ ε, μετριοπαθείς για να μην έχουμε πύριο νίκη. Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες και πρέπει και η κοινωνία να λάβει γνώση της κατάστασης, να ξέρει ακριβώς περί τίνος πρόκειται και να κάνουμε όλοι μια προσπάθεια βιώσιμη, μια προσπάθεια διαρκείας. Δεν πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιούμε συγκυριακή ε, γλώσσα μόνο. Δεν θα αποφέρει αυτό τίποτε. Πρέπει να σας πω ότι είναι πέντε οι βασικοί στόχοι που έχουν τεθεί. δημοσιονομικοί στόχοι, πίστοση, δρομικές μεταρρυθμίσεις, κοινωνικό, στομέας, διοίκηση. Θα πρέπει νομίζω όλα αυτά να γίνουν από κοινού ω προσπάθεια στο δημοσιονομικό επίπεδο θα πρέπει, όπως και στην Ισπανία βέβαια, να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Έχουν ήδη ξεκινήσει, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ε, δεν αρκεί η δημοσιονομική προσαρμογή για την ανάπτυξη. Θα πρέπει να γίνει η δημοσιονομική εξυγίανση και μας έχει δώσει ε, πολύ εύγλωτα μαθήματα η κατάσταση στις Ηνωμένες Δεύτερον, πίστοση, πίστη. Ε, σε ό,τι αφορά την Τραπεζική Ένωση. Πρέπει να ολοκληρωθεί. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη λοιπόν να σκεφτούν. Το μηχανισμό της εξυγίανσης ε, ε, θα τον ε, μεταφέρουν το 2016 και δεν θα πρέπει να δούμε και την πλήρη επιχειρησιακή ισχύ του Ταμείου. Από πότε θα ξεκινήσει, μήπως πρέπει πρώτα να πρικοδευτούν τράπεζες και μετά να καταστεί πλήρως επιχειρησιακός αυτός ο μηχανισμός. Επίσης, πώ οι απώλειες των φορολογουμένων μπορούν να μετριαστούν, τι ευθύνε πρέπει να έχουν οι τράπεζε, θα πρέπει να τα δούμε αυτά. Τρίτο θέμα, δομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να γίνουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό υποστηρίζεται. Αλλά ότι θα πρέπει να είναι προβλέψιμε τι αποφάσει. Και δεν θα πρέπει με την νομοθεσία ε, την αυριανή να καταργείται η σημερινή. Επίσης θα πρέπει να γίνουν επενδύσει να γίνουν για την ανάκαμψη, αλλά αυτό ακόμη δεν έχει συζητηθεί στο κοινωνικό πεδίο. Τα κράτη-μέλη φυσικά και πρέπει να κάνουν μεταρρυθμίσεις, αλλά με προτεραιότητα την απασχόληση, όχι την καταστροφή θέσεων εργασία. Άρα οι μηχανισμοί ευελιξία έχουν στόχο τη διαφύλαξη τη απασχόληση, Άρα το να παίζουμε με μισθού, με μορφέ αλληλεγγύη με ωράριο εργασία δεν είναι σωστό. Επίσης θα πρέπει να εφαρμοστούν και κάποια κατώτατα πρότυπα κοινωνικής προστασίας. Και επίσης, σε ό,τι αφορά τη με τις διοίκησης, και ολοκληρώνω με αυτό, χρειάζεται μια μεγάλη πολιτική συμφωνία και αυτό πρέπει να γίνει. Ζητώ συγγνώμη που σας διέκοψα έτσι απότομα, αλλά υποτίθεται ότι είχατε δύο λεπτά χρόνο. Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο για να μιλήσουμε περισσότερο, αλλά δεν θέλω να είμαι άδικη προς τους υπόλοιπους. Ε, τώρα θα έχουμε την ομιλία του Έντερ Τσεκλούνα που είναι Υπουργός Οικονομικών του Μάλτα και πρώην μέλος της Επιτροπής αυτής. Καλώς επέστρεψες Έντουαρτ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι μιλώ ε, υπό το ρόλο μου ως υπουργός της χώρας μου, όχι το προηγούμενο ρόλο μου όπως, όπως όταν απίθυνα την Ολομέλεια. Ήθελα να μιλήσω λίγο για την ομιμότητα της Τρόικα και το σχετικό ζήτημα. Νομίζω ότι συγχέουμε διάφορα ζητήματα, τα οποία θεωρώ ότι έπρεπε να παραμείνουν ξεχωριστά για να έχει κανείς μια σαφή άποψη του θέματος. Το πρώτο θέμα είναι το κατά πόσο έγιναν λάθη. Και πράγματι έγιναν. Αυτό συνέβη και θα συνέβαινε ανεξάρτητα από το αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα συμμετείχε στην Τρόικα. Εάν ας πούμε οι προβλέψεις ήταν υπερβολικά αισιόδοξε, ότι τα μέτρα λιτότητας δεν θα επηρεάζαν τόσο το ΑΕΠ και ότι οι επενδύσεις δεν θα έπεφταν κατά τόσο μεγάλο ποσοστό ή ότι όλο το ιστορικό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε χώρες που αντιμετώπιζαν σχετικά ζητήματα ήταν επιτυχές επειδή υποτίμησαν το νομισμά του και κατάφεραν να αντισταθμίσουν τα πράγματα μέσω εσωτερικής λιτότητας ε, αλλά ε, ε, εξαγωγών περισσότερων. Αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί όμως στην Ευρωζώνη. Υπήρξαν σημαντικές επιπτώσεις φυσικά στην ανεργία και παρόμοια ζητήματα που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ. Αν έγιναν λάθη, έγιναν διότι υπάρχει έλλειψη τεχνογνωσίας παγκοσμίω για ζητήματα τέτοιου είδου. Οι οικονομολόγοι απλά δεν ε, βρήκαν τα σωστά διορθωτικά μέτρα τη σωστή χρονική στιγμή. Δεν πρέπει λέει, να συγχαίουμε τα λάθη αυτά λοιπόν με το κατά πόσο είχε νομιμότητα ή όχι η Τρόικα. Το δεύτερο είναι το ζήτημα μιας χώρας του Ευρωζώνης που ε, έχασε τον έλεγχο ε, προ όφελο ενό διεθνούς οργανισμού που έχει έδρα τις ΗΠΑ παρά ότι είναι διεθνή οργανισμό. Ε, εδώ μιλάμε για απώλεια ελέγχου μια χρεωμένη χώρα, χώρα κοντά στη χρεοκοπία. Αυτό συμβαίνει παντού. Οποιουσδήποτε άνθρωπο, οικογένεια, επιχείρηση, χώρα πλησιάζει στη χρεοκοπία ή χρεοκοπή, χάνει κάποιον έλεγχο. Έτσι είναι η φύση των πραγμάτων. Χάνει ε, έλεγχο ε, προς όφελος του πιστωτή της τράπεζας που διατίθεται να παρέχει πίστοση εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα θέλει να ανακτήσει τα χρήματα που δάνεισε με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Το ζήτημα λοιπόν της απώλειας ελέγχου δεν έχει να κάνει με νομιμότητα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν υπάρχει δημοκρατία όταν υπάρχουν τόσο σοβαρά ε, οικονομικά προβλήματα. αν πλησιάζετε προσωπικά τη, χροκοπία θα αναμένατε τέτοια πολλή ελέγχου και αυτό μας φέρνει στο ζήτημα της νομότας, της καθεαυτής. Φυσικά, εάν κληθείτε από ένα δικαστήριο, θα προτιμούσετε το δικαστήριο αυτό να βρίσκεται στη χώρα σας, σε ξένη χώρα. Φυσιολογικό είναι. Παρότι η δικαιοσύνη είναι δικαιοσύνη, ε, αλλά αναμένει κανείς ότι τα εθνικά δικαστήρια της χώρα του θα τον κατανοήσουν καλύτερα από ότι ένα ξένο δικαστήριο. Εδώ υπήρχαν λοιπόν κάποιοι όροι και σε περίπτωση τέτοιων όρων προτιμάει κανείς ο θεσμός αυτός, δηλαδή η Τρόκα, να βρίσκεται πιο κοντά στη χώρα μας, δεν είναι πιο ευρωπαϊκή από από τη διεθνής ε, υπό τέτοιε περιστάσεις. Πρέπει να διαχωρίσουμε όλα αυτά τα σημεία μεταξύ τους, ώστε να μπορέσουμε να συμπεράνουμε κατά πόσο υπήρχε νομιμότητα ή όχι. Αλλά ξέρετε, όταν λαμβάνει κάποιες συστάσει, αυτές πρέπει να γίνονται κατανοητές από τους ανθρώπους. Ναι, σύμφωνο, έπρεπε να υπήρχε μεγαλύτερη νομιμότητα νομότα, τουλάχιστον όπως την αντιλαμβάνονται οι κάτοικοι των χωρών, των χωρών αυτών που εντάσσονται στο πρόγραμμα αναπροσαρμογή. Ευχαριστώ, Εντουάρντα, από την Κροατία, από την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Έχουμε το Ιβάνα Μάλετσο. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ η Κροατία βρίσκεται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό για μένα που είμαι πρόσωπο της Κροατίας είναι να δω τι μηχανισμοί υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, το οποίο μας επιτρέπει να λαμβάνουμε μακροπρόθεσμα διαρθρωτικά μέτρα, τα οποία θα μας επιτρέψουν να απαντήσουμε στο ερώτημα πώς μπορούμε να αυξήσουμε τις επενδύσεις, πώς μπορούμε να μειώσουμε την ανεργία. Όμως, τις απαντήσεις τις ξέρουμε όλοι σε αυτά τα ερωτήματα. Το πρόβλημα αλλού έγκυται. Πώς θα τις εφαρμόσουμε τις λύσεις. Εάν θέλουμε να αυξήσουμε τις επενδύσεις, πρέπει να είναι ασφαλές το επενδυτικό κλίμα. Εάν θέλουμε να αυξήσουμε τις εξαγωγές, πρέπει να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας. Πρέπει επίσης να βρούμε και άλλους πόρους, ε, να υπάρχουν και άλλες πηγές χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις. Άρα, γνωρίζουμε τις απαντήσεις, αλλά δεν ξέρουμε πώς να τις εφαρμόσουμε στην πράξη. Εξού και είναι ανάγκη ε, να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή εμπειριών, όπως σήμερα διότι μιλάμε για την διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε τάχιστα τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που θα μπορούσαν να έχουν άμεσο αντίκτυπο. Και ξέρετε, κάθε μέτρο μπορεί να είναι θετικό, μπορεί να είναι όμως και αρνητικό. Παραδείγματο χάρη, θέλουμε να μειώσουμε ε, τους μισθούς στο δημόσιο τομέα. Γιατί έτσι μειώνεται σχεδόν αυτομάτως το έλλειμμα. Όμως, με τον τρόπο αυτό, κατεβαίνουν, πέφτουν και οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα. Οπότε οι επιχειρήσεις γίνονται λιγότερο ανταγωνιστικές. Και αν μειώσουμε τους μισθούς κάτω από ένα αποδεκτό εύλογο επίπεδο, μειώνεται ο αριθμό των υπαλλήλων, των εργαζομένων και αντί να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, μειώνεται. Υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα λοιπόν Πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε όλα αυτά τα μέτρα να τα εφαρμόσουμε στην πράξη, ώστε να δώσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Εγώ πιστεύω ότι το παράδειγμα της Ολλανδίας είναι καλό. Πρέπει να συνεργαστούμε με όλους τους κλάδους της κοινωνίας για να προωθήσουμε αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις και για να ενισχύσουμε τη διοίκηση με την αποτελεσματική αποκέντρωση. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε τώρα από ένα άλλο μέλος της Επιτροπής Εικόνα από την Ισπανία, ε, πρόεδρος Παύλος Ζέλβα. Σαρών. Σε ευχαριστώ Σάρων. Εγώ χαίρομαι που έχει αλλάξει σελίδα αυτή η ψευδοσυζήτηση μεταξύ λιτότητας ε, ή ανάπτυξης. Και εγώ καταλαβαίνω ότι συμφωνούμε όλοι ότι φυσικά και πρέπει να είναι ε, εξυγιασμένοι λογαριασμοί για να έχουμε οικονομική ανάπτυξη, να έχουμε εξυγίανση. Ο Πέτρος Σόρα είπε ότι πρέπει να βρούμε την κατάλληλη στιγμή. Συμφωνώ. Και νομίζω ότι αυτό έκανε η Ισπανική κυβέρνηση που κατάφερε στη θητεία αυτή μέσα σε δύο-τρία χρόνια να έχουμε άλλα δύο-τρία χρόνια στη διάθεσή μας για να ε, ικανοποιήσουμε τους στόχους ε, του ελλείμματος και αυτό είναι αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης ε, που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον στην Ισπανία τη αξιοπιστία που εμπνέουμε. Πρέπει τώρα όμω να προωθήσουμε την ανάπτυξη. Και κάτι με δύο είναι τα θέματα προτεραιότητα. Μεταρρυθμίσει, όπω είπαμε και στη συζήτηση τη χθεσινή, να συνεχίσουμε τη μεταρρυθμιστική ορμή, όπω εμεί, όπω και άλλα πολλά κράτη-μέλη τη Ένωση και η πλέον διστακτική και επιφυλακτική ή να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν να προωθούν τις μεταρρυθμίσεις αυτές. Κάτι άλλο που συζητήσαμε επίση χθε είναι ότι οι επιχειρήσει και οι δύο μικρομεσαίε επιχειρήσει πρέπει να έχουν πρόσβαση στην πίστη, σε δάνεια, με όρου αντίστοιχου αυτών τη Ευρωζώνη. Αυτή είναι μεγάλη πρόκληση και για μα μεγάλη πρόκληση για φέτο. Γιατί η ΜΜΕ θα είναι μοχλός θα είναι οι ε, πρωταγωνίστρες της οικονομικής ανάπτυξης. Για να γίνει αυτό όμως δεν είναι αποκλειστικά εθνική λύση, αλλά ευρωπαϊκή. Γιατί οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι κατακαιρματισμένες και γι' αυτό τα κράτη-μέλη, η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να ενεργούν με τον ίδιο τρόπο. Ελπίζω αυτή η ορχήστρα που τη συναπαρτίζουν όλοι αυτοί να μην είναι παράφωνοι και να αρχίσουν να ρέουν οι πόροι. Διότι, όπως είπε και ένας συνάδελφος, ε, βοηθάει και η Τραπεζική Ένωση. Αλλά αυτό μακροπρόθεσμα, μέσο μακροπρόθεσμα, βράχη πρόθεσμα, χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Χρειαζόμαστε τη μεγαλύτερη συμμετοχή της Τράπεζας Επενδύσεων και της Κεντρικής Τράπεζας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Thank Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα έχουμε ένα γερουσιαστή από την Επιτροπή Προπολογισμού της Ιταλίας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι εχθές και σήμερα είπαμε ότι θέλουμε να ξεκινήσει μια νέα φάση στην Ευρώπη που να καταλήξει στην οικονομική ανάπτυξη. Για να υπάρχει λοιπόν οικονομική ανάπτυξη χρειαζόμαστε διαρθρωτικές αλλαγές. Αυτό είπαμε. Εγώ πιστεύω ότι για να αποφύγουμε και άλλες απογοητεύσεις στο μέλλον θα πρέπει να διευκρινίσουμε την κατάσταση ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αρκετοί αμφισβητούν την ανάγκη ύπαρξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην Ευρώπη. Ε, πρέπει, λένε, να υπάρξει ταχύτατη ανάπτυξη και αυτό μεταξύ άλλων απαιτεί περισσότερο ευέλικτες και ανταγωνιστικές ε, αγορές. Πρέπει όμως να προσθέσουμε θέσουμε ότι οι διαφορετικές μεταρρυθμίσει μόνες τους δεν θα οδηγήσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Τουν αντίον βράχτεσμα τέτοιου είδου ε, μεταρρυθμίσεις ε, θα μειώσουν περαιτέρω τη ζήτηση. Έτσι λοιπόν οι διαφορετικές μεταρρυθμίσεις ε, μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα μέσα από δύο παράλληλα κανάλια. Το ένα είναι η ζήτηση που ε, έχει συνδυαστεί με την παραγωγικότητα. Χρειαζόμαστε πάντως και τις δύο διαδικασίες παράλληλα για να επιτύχουμε οικονομική ανάπτυξη. Για να δούμε ε, τι μπορεί να συμβεί αν η συνολική ζήτηση περιοριστεί όπως σημαίνει τώρα στην περιφέρεια της Ευρώπης. Η, ε, το αγοραστικό το ανθρώπινο δυναμικό δεν θα λειτουργεί αποτελεσματικά, άρα δηλαδή την εργασία την ε, αφαιρούμε από την χαμαλή παραγωγικότητα και τέλος ε, η ανεργία επιδεινώνεται. Άρα δηλαδή Νομίζω ότι θα πρέπει με απόλυτη σοφήνεια να τανίσουμε ότι η στρατηγική για να έχουμε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η δυνατότητα αυτή είναι ή πρέπει να βασίζεται σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αφενός αλλά αφετέρου και σε τρία άλλα βασικά στοιχεία που αφορούν στη συνολική ζήτηση. Δηλαδή συμμετρική μακροοικονομική προσαρμογή ε, σε σχέση με το έλλειμμα και το πλεόνασμα, μια αποτελεσματική τραπεζική ένωση, αυτό είναι καθοριστική σημασία, και το τρίτο, χρειαζόμαστε επενδύσεις επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και σε επίπεδο κρατών μελών. Δεν μπορούμε να περιζόμαστε μόνο στις διαρθρωτικέ αλλαγές. Υπάρχουν πάρα πολλές αμφιβολίες για το κατά πόσον στο τέλος ε, θα έχουμε παραγωγικό τομέα. Δεν θα, είναι ε, αύξηση, δεν θα υπάρξει αύξηση της παραγωγικότητας, του αντίον θα υπάρξει αύξηση της ανεργίας. Ευχαριστούμε πολύ τώρα η Μαρία Τάισεν, άλλο μέλος της ΕΚΟΝ από το Βέλγιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όταν μιλάμε για δημοσιονομική εξυγίανση και για ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ε, συχνά αναφερόμαστε και σε εθνική κυριαρχία. Πολύ το ανέφεραν σήμερα συνάδελφοι. Γνωρίζω επίσης ότι πολλές χώρες ε, καλούνται να λάβουν δύσκολες αποφάσεις και ότι η πίεση που απορρέει από τις ε, ευρωπαϊκές συμφωνίες ε, είναι πολύ ψηλή για τα κράτη-μέλη. Οι προσπάθειες που ζητούνται είναι ευρείας κλίμακας συχνά. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να παρακαλέσω και να παροτρύνω τους εθνικούς βουλευτές να περάσουν το εξής μήνυμα Ας μην διακομωδούμε την κατάσταση. Ας μην ε, κάνουμε τους ανθρώπους να νομίζουν ότι όλες αυτές οι ευρωπαϊκές αποφάσεις επιβάλλονται στους πολίτες ε, ως αν η Ευρώπη να ήταν ε, ένας ξένος παράγοντας που επιβάλλει κάτι στις χώρες αυτές. Η Ευρώπη δεν είναι το εξωτερικό, είναι η κοινή μας χώρα. Μιλάμε για ευρωπαϊκές αποφάσεις στις διάφορες πρωτεύουσες και τίθεται και το ζήτημα της κυριαρχίας. Ε, ε, έχουμε μια κοινή κυριαρχία, κοινή εθνική κυριαρχία που βασίζεται στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Συνδυάζουμε τις δυνάμεις μας, τα πλεονεκτήματά μας ε, για να δράσουμε πιο στοχευμένα, πιο αποτελεσματικά. Και αυτό επιτρέπει να περνάμε και καλύτερα τι ευρωπαϊκές Συμφωνίε του πληθυσμού μα Να υπενθυμίσω λοιπόν στου συναδέλφου, μην λέτε η Ευρώπη μα υποχρεώνει. Γιατί αυτό δυσκολεύει την αποδοχή από του πολίτε ε, τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ζητήστε κατανόηση. Εξηγήστε στου πολίτε. ότι σίγουρα ναι αυτέ οι αποφάσει προέρχονται από την Ευρώπη αλλά είναι ωφέλιμε. Δεν είναι εύκολο κάποια χώρα να λαμβάνει τόσο ευαίσθητε αποφάσει. Μερικέ φορέ είναι υπερβολικά ευαίσθητα τα ζητήματα και δύσκολες οι αποφάσεις, μερικές φορές ε, με συνέπειες μακροπρόθεσμες. Πρέπει να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι η Ευρώπη βρίσκεται εδώ για να μας βοηθήσει όλους να παραμείνουμε σε έναν δρόμο ευημερίας. Φυσικά και πρέπει από την άλλη πλευρά να αξιολογούμε, να διορθώνουμε, να επικρίνουμε τις πολιτικές ε, που ακολουθούμε, να λαμβάνουμε υπόψη τα χρονοδιαγράμματα και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά σας παρακαλώ, ας μην τα κάνουμε όλα αυτά ε, έχοντας την Ευρώπη σαν να έπρεπε για εχθρός ε, των κρατών μελών σαν να έχει δίκιο είτε ο ένας είτε ο άλλος. Είμαστε όλοι μαζί, μια ομάδα. Δεν υπάρχει μάχη μεταξύ χωρών που είναι αλληλέγγυες. Δεν υπάρχουν αλληλέγγυες και μη αλληλέγγυες χώρες, οι χώρες που υποφελούνται της αλληλεγγύης. Είναι κοινή η αλληλεγγύη, οι στόχοι είναι κονοί, όλα είναι κοινά και πρέπει να παραμένουν κοινά για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να έχουμε ε, ανάπτυξη για μεγάλο, για πολλά χρόνια. Αυτά ήθελα να πω κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η έννοια της εθνικής κυριαρχίας πρέπει να αξιολογηθεί με την πραγματική της αξία και πιστεύω ότι κάθε διοικητικός οργανισμός στην Ευρώπη πρέπει να αναλαμβάνει τις δικές του ευθύνες. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουν μείνει άλλε κάρτε από την αίθουσα. Να επανέλθω λοιπόν στα μέλη που ε, καθίξαν τη συζήτησή μα ε, Δίνω το λόγο στην κόρη. Θέλετε να ξαναπάρει το λόγο, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση πράγματι. υπάρχουν κάποια σημεία επαφή. Όλοι συμφωνούν ότι θέλουμε μεταρρυθμίσει. Όλοι συμφωνούν ότι αυτέ θα είναι επώδυνε και ότι θα χρειαστεί να εξηγηθεί η ωφελημότητα των μεταρρυθμίσεων αυτών και ότι αυτό είναι ένα μήνυμα πρέπει να διαβάσουμε στους πολίτες μας. Πιστεύω επίσης ότι διαπιστώνουμε όλοι μαζί ότι αυτό που συμβαίνει σε μία χώρα μπορεί να έχει εντυπωσιακά σημαντικές επιπτώσεις σε μια άλλη χώρα. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε αναγκασμένοι να προσέχουμε ιδιαίτερα τι κάνουμε. Και για να ολοκληρώσω κυρία Πρόεδρε, να κάνω μια έκκληση, να προβληματιστούμε λίγο, να αξιολογήσουμε τα μέσα από τους μηχανισμούς που έχουμε δημιουργήσει, να μελετήσουμε την αποτελεσματικότητά τους, την απόδοση αυτών των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και να δούμε πώς θα προσεγγίσουμε αυτό το φαινόμενο των μεταρρυθμίσεων. Ε, καλό είναι φυσικά να ανταλλάσσουμε βέλτιστες πρακτικές. Για παράδειγμα, το ελεκτικό συνέδριο ε, των κατοχωρών ε, εξετάζει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται σε θέματα δημοσίων οικονομικών και προπολογισμού και πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να αποφεληθούμε από την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό είναι και ο σκοπό ε, αυτή εδώ τη διάσκεψη. Ε, συζήτηση μεταξύ των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να δράξουμε αυτή την ευκαιρία, να ανταλλάξουμε απόψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σας ευχαριστώ πολύ. Η συζήτηση αυτή με ικανοποίησε και με εμπλούτησε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι όταν μιλάμε για καλές πρακτικές είναι πολύ σημαντικό να διδασκόμαστε από το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Να βλέπουμε τι ενέργειες γίνονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να εφαρμόσουμε μέτρα που θα μας ωφελήσουν και εμάς. Όμως, εξίσου σημαντικό είναι να υπογραμμίσουμε ότι καλές πρακτικές σήμερα είναι απαραίτητες διότι αυτό που κάνει μία χώρα μέλος επηρεάζει και άλλες χώρες μέλη. Πιστεύω ότι καλές πρακτικές δεν είναι μόνο μία μέθοδος εκμάθησης, αν θέλετε, αλλά είναι ανάγκη για να τα πάμε όλοι καλύτερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ευρώ, για τις χώρες μέλη συνεπάγονται ανάπτυξη και όχι απλά αναλογική. Θα πάει πιο καλά ε, η κατάσταση, αλλά μόνο εάν ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση και τα πηγαίνουμε καλά. Στη δική μου χώρα πιστεύουμε ότι οι ιδιαιτερότητες των χωρών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να συνδυάζονται με συνεκτικές, συνεπείς πολιτικές που θα τις εφαρμόσουν όλοι. Και από αυτήν την έννοια θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι ναι δεν πρέπει να απολέσουμε την κυριαρχία μας, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να οδηγήσει τις χώρες σε ένα μονοπάτι ώστε οι μένουν να μην θέτουν σε κίνδυνο τις δε. Κατ' εμέ αυτό είναι ένα δίδαγμα που μπορούμε να αντλήσουμε από την κρίση. Νομίζω ότι η κρίση κατέδειξε την ανάγκη χωρίς, επαναλαμβάνω, απώλεια κυριαρχίας, την ανάγκη συντονισμού των οικονομικών πολιτικών των χωρών. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι από το Ισπανικό Κοινοβούλιο ήρθα στην Ευρώπη, σας μετέφερα τις συζητήσεις που έχουμε στο Ισπανικό Κοινοβούλιο εξήγησε και ο κύριος Σάντσεφ Πρεσέδο μερικά πράγματα σε ό,τι αφορά τα στοιχεία για το δημόσιο έλλειμμα. Είδαμε και ο κύριος Σάουρα είπε τα σχετικά. Ίσως όλες αυτές οι υποθέσεις που ακούμε και τα στοιχεία ουσιαστικά, τα νούμερα δείχνουν την πραγματικότητα και αυτά τα νούμερα που έχουμε στην Ισπανία τα επιβεβαιώνει και η Eurostat, τα επιβεβαιώνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βέβαια και τα ισπανικά κόμματα συζητάμε μεταξύ μα και νομίζω ότι σήμερα μπορώ να σα πω και φαντάζομαι θα συμφωνήσουν οι συναδελφοί μου ότι τα δύο τελευταία χρόνια η Ισπανία είναι μια περίπτωση επιτυχία. Δηλαδή εξερχόμαστε, βγαίνουμε από αυτή την κατάσταση. Τυχαίο θα πει ένα συνάδελφο ίσως από την αντιπολίτευση. Όχι, δεν είναι τυχαίο θα πω εγώ, είναι γιατί κάνουμε καλά τα πράγματα. Ε, thank ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν βλέπω να επιθυμεί κάποιος άλλος να λάβει το λόγο. Δεν ξέρω μήπως επιθυμεί κάποιος ε, να λάβει το λόγο. Κάποια από τα θέματα που τέθησαν ε, μας απασχολούν πάρα πολύ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή συζητάμε για το πώς είναι δυνατόν να επιτευχθεί η ε, συμμετρική προσαρμογή. Αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα επίμεχο, αλλά κάπως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και νομίζω ότι πολύ σωστά ελέγχθη προηγουμένως ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε όλοι οι πιστωτές προφανώς και επιβάλλουν όρους. Αυτό τον έφερε ο κύριος Σικλούνα και επίσης ε, πρέπει να πούμε ότι ορισμένα κράτη-μέλη αναζητούν ε, τους τρόπους, τις δυνατότητες ε, για να γίνει κατανοητό ότι τα αφορούν άμεσα αυτά τα θέματα διότι αλλιώς δεν μπορεί κανείς να προβεί σε σημαντικές αλλαγές αν δεν οδηγεί στους πολίτες στο να κατανοήσουν ότι όλα αυτά τα θέματα τους αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει αυτά να τα χειριζόμαστε μόνοι μας και όχι να καταφεύγουμε σε βοήθεια από το εξωτερικό. Στις 11.30 θα ξεκινήσει η επόμενη συνεδρία. Μπορούμε να έχουμε ε, ένα διάλειμμα για λίγα λεπτά και στις 11.30 θα έχουμε την καταληκτική συνεδρία όπου θα συμμετέχουν και συνάδελφοι από την Επιτροπή Απασχόλησης και Προϋπολογισμού. Και όσοι δεν έχετε ενημερωθεί, να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέριψε την ε, προσφυγή του Ρωμανού Βασιλείου για το short selling. Ε, ακόμα δεν έχω να σας πω λεπτομέρειες. Ε, αυτά είναι τα νέα της τελευταίας στιγμής. Πριν από τρία τέταρτα εκδόθηκε η απόφαση και απλά σας ανέφερα. Θα επανέλθουμε στις 11.30.